And... Καλή σας μέρα. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Ξεκινάμε το σημείο 15 της ημερησίας διάταξης. Παρουσίαση της μελέτης για το ποινικό δικονομικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως θα θυμάστε το άρθρο 82 της ε, συνθήκης περί αμοιβές αναγνώσεις σε ποινικά θέματα αποτελεί νομική βάση για την εναρμόνιση ορισμένων δικονομικών πτυχών, δικαιώματα των υπόπτων, θυμάτων ε, και κατηγορουμένων. Αυτό είναι σημαντικό για την αμοιβαία αναγνώριση σε ποινικά ζητήματα. Έχουμε αρκετή εμπειρία από το ένταλμα σύλληψης ε, και από αυτό προκύπτει ότι χρειάζεται διεύρυνση των κανόνων, ε, της εναρμόνισης των κανόνων. Το θέμα είναι ευαίσθητο ε, και πολύ συχνά υφίστανται εθνικές, νομικές και πολλές φορές και συνταγματικές, συνταγματικά προβλήματα. Η Υπάρχει και μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την οποία θα μιλήσουμε και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ειδοποίησης για Υπόπτους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία επηρεάζουν τους κανόνες αυτούς. Η εναρμόνιση επίσης λαμβάνει η χώρα σε ό,τι αφορά το παραδεκτό των τεκμηρίων για συγκεκριμένα ανακριτικά, συγκεκριμένες ανακριτικές διαδικασίες. Θα μας μιλήσουν δύο εμπειρογνώμονες πριν δώσουμε το λόγο στα μέλη. Καταρχήν έχουμε την καθηγήτρια Αν Βέιμπεργκ και την κυρία Έλοντι Σέλερ, τις οποίες καλωσορίζουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τους ειδικού και μετά θα συζητήσουμε και μεταξύ μας. Καθηγήτρια Βέμπερ, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τιμή και χαρά για την Σελέ και για μένα να σας παρουσιάσουμε εν συντομία τη μελέτη μας. Αν επιτρέπετε, μερικά λόγια να σας υπενθυμίσουμε το ιστορικό της υπόθεσης. Εδώ και 20 περίπου χρόνια ε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εμβέας αναγνώρισης για ποινικέ υποθέσεις. Μια διαδικασία που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, δικαιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών. Πολλά έχουν λεχθεί και γραφεί για την αμοιβαία μισθοσύνη. Πολλές φορές έχει γίνει έκκληση η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση προκειμένου ε, να συγκλίνουν ε, οι δικονομικές διαδικασίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Η θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας αποτέλεσε ορόσημο σε αυτή την προσπάθεια. αποτελεί μία κίνηση προς την προσέγγιση με βάση τις αρχές και γι' αυτό το λόγο είχαμε ε, μία σειρά δικαιωμάτων όπως για παράδειγμα δικαιώματα ε, στην μετάφραση και την ε, διερμηνία, παρουσία δικηγόρου ή νομικής συνδρομής, ε, δικαιώματα προστασίας των θυμάτων και, των, και προστασία των παιδιών στόχος του συστήματος, ε, στόχος της μελέτης ε, τη δική μας ήταν να ξεπεράσουμε αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει γίνει η διεναρμόνιση. Θεωρούμε ότι είναι πρόωρο να ζητήσουμε μια αναθεώρηση των 7 οδηγιών που έχουν υιοθετηθεί. Οπότε η μελέτη επικεντρώθηκε στο να εντοπίσει άλλους τομείς ε, δικονομικών διαδικασιών στους οποίους οι διαφορές στους εθνικούς νόμους επηρεάζει την διασυνοριακή συνεργασία ή την συνεργασία, την διαπραγμάτευση γνώμη και την υιοθέτηση νέων νομοθετικών κυμάτων που, κειμένων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, ακολουθήσαμε μια συγκριτική νομική προσέγγιση επί τη βάση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εννέα κρατών μελών που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές παραδόσεις και που γεωγραφικά είναι ε, ποικίλε. Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, κάτω χώρες, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Ήταν αυτές οι εννιά χώρες. Η ανάλυση βασίστηκε σε έρευνα που έγινε στο γραφείο, σε, επίσης βασίστηκε σε εννέα εθνικές εκθέσεις και σε συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες στις, ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς, δίκτυα και σε, με εθνικούς εμπειρογνώμονες. Ως αποτέλεσμα εντοπίσαμε εννέα τομείς στους οποίους οι διαφορές ανάμεσα στις ε, εθνικές ε, ποινικέ διαδικασίες αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης και της, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η λέξη εμπόδιο ε, πρέπει να ειδωθεί με ευρύ τρόπο και πρακτικά στη συνεργασία αλλά και ως εμπόδιο στην άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων. Οι εννέα είναι οι εξής. Πρώτον, ανακριτικά μέτρα. Δεύτερον, παραδεκτό των τεκμήριων. Τρίτον, η ποιότητα των ε, μέσων που χρησιμοποιούνται. Ε, κράτηση πρώτης δίκης ερημοδικία, αποζημιώσεις για ε, αδική κράτηση, αποζημιώσεις για τα θύματα και προστατευτικά μέτρα, μέτρα προστασίας των θυμάτων. Πριν εξετάσουμε ένα προς ένα αυτούς τους τομείς, να σας πω ότι Είχαμε πολλές προκλήσεις ε, και σε ό,τι αφορά το εύρος ε, όσο και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ε, οπότε μην θεωρήσετε ότι όλα όσα λέμε έχουν εξαντλήσει το ζήτημα. Η Ελλοντή θα, θα συνεχίσει με την παρουσίαση με τους πρώτους τρεις τομείς. Καλή σας μέρα. Καταρχήν εξετάσαμε τα ανακριτικά μέτρα. Υπάρχει πολύ ερευνητική διαδικασία, ε, αλλά υπάρχει και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί τεκμηρίων. Η πρώτη διαφορά που, ανακαλύψαμε, που εντοπίσαμε, ήταν ο βαθμός εμπλοκής των διοικητικών αρχών. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη βασίζονται στην ε, συνεισφορά ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Ε, επίσης, ε, η διαφορά ανάμεσα στα νομικά συστήματα που κάποια δίνουν σημασία, πιο πολύ σημασία στον εισαγγελέα, αλλά στον ανακριτή, αλλά δεν έχουν ανακριτή καθόλου. Δεν υπάρχει κοινό κατόφλι για την εκκίνηση μιας ανάκρισης, ούτε έχουμε κοινέ διαδικασίες για την ε, α, αίτηση άδεια. Έχουμε επίσης πολλές φορές πολλές διαφορετικές εθνικές αρμόδιες αρχές. και επίσης μερικές φορές ε, προβλέπεται η παρεμβολή και μη δικαστικών. Οι διαδικασίες επίσης πολλές φορές είναι πολύ περίπλοκες. Ε, ε, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από μια, ένα κεντρικό γραφείο έχουμε καταλήξει μετά από πολλές διαπραγματεύσεις σε, σε αποκέντρωση και αυτό δημιουργεί επίσης προβλήματα. Ε, είναι πολλές ε, φορές επίση πολύ δύσκολο να εντοπιστεί στα κράτη-μέλη ε, το, η αρμόδια αρχή προκειμένου να σταλεί έτοιμα έρευνας. Σε ό,τι αφορά το, το, το διοικητικό βάχθος, δεδομένου ότι έχουμε πολλές φορές και διοικητικό και ποινικό δίκαιο το οποίο εμπλέκεται σε διάφορε υποθέσει, αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί πολλές φορές οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί, το διοικητικό δίκαιο ή το ποινικό δίκαιο και οι αντίστοιχες ε, ε, ρήτρες προστασίας. Ε, στο ποινικό δίκαιο οι ρήτρες αυτές είναι πιο ισχυρές, για παράδειγμα. Μετά, το αποδεκτό των τεκμήριων. Εστιάσαμε σε τεκμήρια τα οποία έχουν συλλεχθεί νομίμως. Γι' αυτά δεν υπάρχει κανόνας τις Ευρωπαϊκή Ένωσης. Τα συστήματα παραδεκτού είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ κρατών μελών. Μερικά κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένου κανόνε αποκλεισμού, για παράδειγμα, ε, τεκμήρια τα οποία έχουν συλλεχθεί με ε, βασανιστήρια ξερούνται αυτόματα. Ενώ άλλα κράτη-μέλη βασίζονται στη διακριτική ευχαίρεια του δικαστή. Ο δικαστή θα αποφασίσει αν τα τεκμήρια θα γίνουν δεκτά ή όχι. Σε ό,τι αφορά την, τις επιπτώσει, επιπτώσεις, έχουμε ένα σύστημα δύο επιπέδων. Ε, για παράδειγμα, για τις, ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις κοινές ομάδες έρευνα, ε, εφαρμόζεται το δίκαιο του εκτελώντος κράτους μέλους ενώ για την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας ε, εφαρμόζεται το δίκαιο της, του ετούντος κράτου μέλους. Αυτό περιπλέκει πολύ τα πράγματα. Για παράδειγμα, στην οδηγία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας ε, ο, το, το ετών ε, κράτος ε, εφαρμόζονται οι κανόνες του ετούντος ε, κράτους μέλους, οπότε το εκτελών κράτος μέλος δεν ξέρει ποιους κανόνες να εφαρμόσει ακριβώς. Αυτό μας το υπέδειξαν ε, ε, στη συνεντεύξεις Είναι πάρα πολύ προβληματικό θέμα. Ο, ο κατηγορούμενος, για παράδειγμα, αν θέλει να αμφισβητήσει ένα τεκμήριο το οποίο έχει συλλεχθεί αλλού, ε, δεν ξέρει πού έχει συλλεχθεί. Και αυτό είναι πολύ ε, σημαντικό διότι ε, προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά, ισότητα των μέσων σε διασυνοριακές ανακρίσεις. Δεν θα πρέπει ο κατηγορούμενος να βρίσκεται σε υποδέστερη θέση. Αν όμως θέλει να εφαρμόσει, τη, να κάνει τη δική του έρευνα ε, για να βρει τεκμήρια που τον αθώνουν, θα αντιμετωπίσει πολλά πρακτικά προβλήματα όπως η γλώσσα και άλλα. Θα μιλήσουμε αργότερα για τους όρους και τις σύνθηκες κράτησης. Περνάμε τώρα στην ε, στο τέταρτο θέμα μας ανησυχεί, το οποίο αφορά την ε, κράτηση πρώτης δείξης. Τα καθιστώτα της ε, προφυλάξης διαφέρουν ε, κατά πολύ. Διαφέρουν όσον αφορά την διάρκεια της κράτησης. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ένα μέγιστο τέτοιο όριο, το οποίο ποικίλει. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει κάποιο όριο, αλλά εφαρμόζονται χρονικά όρια σε κάθε φάση της ε, προφυλαξής και υπάρχει ένα σύστημα εξέτασης από τα δικαστήρια. Επίσης αποκλίνουν κατά πολύ τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται για να υπάρξει κάποια προφυλάξη. Και αυτό το οποίο διαφέρει πολύ στα εθνικά συστήματα είναι το όριο, το επίπεδο της υποψίας ε, το οποίο απαιτείται για να υπάρξει μια προφυλάκηση. Τέλος, έχουμε την φύση των εναλλακτικών στην ε, κράτηση μεταξύ των κρατών μελών. Οι διαφορές αυτές επηρεάζουν σοβαρά την διασυνοριακή συνεργασία. Τα εμπόδια στην ε, αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη προκύπτουν άμεσα από την διαφορετική ερμηνεία των καθεστώτων κράτησης και ειδικά από το διαφορετικό επίπεδο υποψία στο οποίο απαιτείται. Βεβαίως ε, μια μεγάλη περίοδος ε, προφυλάξης ε, σημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο δεν γίνεται εκτός σε κάποια κράτη-μέλη, τα οποία αρνούνται να εκτελέσουν αιτήματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό το οποίο θεωρούν υπερβολική χρήση της ε, κράτησης. Οι διαφορές επίσης στις εναλλακτικές της ε, κράτησης επίσης εμποδίζουν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Το θέμα αυτό λοιπόν σημαίνει ότι συχνά υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ των κρατών μελών. Πέραν λοιπόν από την μη χρήση αυτού του μέσου έχουμε και την έλλειψη επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των αρχών. Τώρα θα περάσω στον πέμπτο τομέα που μας ανησυχεί και είναι οι συνθήκες της ε, κράτησης μετά από αυτήν την πολύ γνωστή απόφαση του δικαστηρίου Αρανιόζιεν και Καλντεράρου. Θα γνωρίζετε βεβαίως ε, την απόφαση αυτή του Απριλίου του 2016. Όπως ε, ξέρετε η απόφαση αυτή έδωσε το πράσινο φως στις ε, αρχές ε, του εκτελούντος ε, μέλους να αρνηθούν την παράδοση αν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι το άτομο θα εκτεθεί σε απάνθρωπη και ταπεινωτική συμπεριφορά. Για να γίνει αυτή η αξιολόγηση, οι εθνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες από την αρχή η οποία έχει εκδώσει το αίτημα όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης είχαμε και την απόφαση της 25ης Ιουλίου 2018 στην λεγόμενη υπόθεση ML. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το είδος των πηγών για την αξιολόγηση, για το εάν θα πρέπει να παραδοθεί κάποιος σε άλλο κράτος, τα αιτήματα για πληροφορίες τα οποία αποστέλλονται στα κράτη τα οποία εκδίδουν τα αιτήματα επίσης διαφέρουν. Διαφέρει ο βαθμός λεπτομέρειας Καμιά φορά οι αρχές οι οποίες εκτελούν το αίτημα πηγαίνουν παραπέρα από αυτό και για να υπάρξει παράδοση του κρατουμένου ζητάνε κάποιες εγγυήσει ή διαβεβαιώσεις που παραδείγματο χάρη μπορεί να αφορούν την παροχή ε, ατομικού κέλιου στον ε, κρατούμενο. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου βεβαίως ε, είναι καλοδεχόμενη, αλλά οι πρακτικές που αναφέραμε έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αμοιβαία αναγνώριση και την εμπιστοσύνη. Και αυτές ξεκινάνε από καθυστερήσεις μέχρι και άρνηση εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα με την Γερμανία. Μία υπόθεση είχε πάει στο ανώτατο δικαστήριο το 2014 και αφορούσε ακριβώς τις συνθήκες ε, κράτησης ε, στην περίπτωση εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού εντάλματος ε, σύλληψης από τις 40 υποθέσεις του 2016. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος πόλωσης μεταξύ των κρατών μελών με καλές και κακές φυλακές. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος επιλογής φυλακών από τους κατηγορούμενους το σύστημα αυτό παροχής εγγυήσεων ή διαβεβαιώσεων επίσης έχει κάποιες ανησυχίες, παραδείγματο χάρη οι διαφορές ε, στην αντιμετώπιση που δημιουργεί το σύστημα για άτομα που εμπλέκονται σε διασυνοριακές υποθέσεις και αυτά τα οποία εμπλέκονται σε καθαρά εθνικές υποθέσεις ε, που δεν έχουν τέτοιες εγγύησεις. Ένα άλλο θέμα επίσης μας ανησυχεί είναι το ότι είναι πολύ δυσκίνητο το σύστημα αυτό των εγγύσεων σε μεγάλη κλίμακα. Είναι αδύνατο για χώρες με κακές συνθήκες κράτησης να εγγυηθούν ατομικά κελιά σε μεγάλη κλίμακα. Πέρα από αυτές τις ανησυχίες, το θέμα των συνθήκων κράτησης πράγματι επηρεάζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη εντός της Ένωσης και όχι μόνο στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, αλλά στην περίπτωση όλων των μηχανισμών συνεργασίας που αφορούν την κράτηση και στο πλαίσιο της απόφασης πλαισίου για την μεταφορά κρατουμένων. Το έκτο θέμα που ε, θεωρήσαμε ανησυχητικό είναι η αποζημίωση για άδικη κράτηση στις ε, διεθνείς ε, αυτές διαδικασίες αλλά σας παραπέμπουμε εδώ στην μελέτη, δεν υπάρχει χρόνος τώρα να ασχοληθούμε με αυτό. Το έβδομο ε, σημείο ανησυχίας είναι οι δίκες ερήμην. Εδώ πέρα υπάρχουν σοβαρές ε, διαφορές που δημιουργούν διάφορα εμπόδια στην διασυνοριακή συνεργασία, αλλά αφού ο χρόνος ε, πιέζει θα το προσπεράσουμε και αυτό. Και σας παραπέμπουμε στην μελέτη και τώρα θα δώσω τον λόγο στην Ελοντή για τα δύο τελευταία σημεία ανησυχίας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο σημεία έχουν μείνει ε, που αφορούν τα δικαιώματα των θυμάτων. Υπήρχε τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, εν μέρη και λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα πολλές ε, ανισορροπίες όσον αφορά την αντιμετώπιση των θυμάτων. Η αποζημίωση των θυμάτων είναι ένα από αυτά. Υπήρχε μια οδηγία του 2004 για την διασυνοριακή αποζημίωση, αλλά η οδηγία δεν προβλέπει κανενός είδους εναρμόνιση όσον αφορά και προθεσμίες για να υπάρξει ένα σύστημα εναρμόνισης. Οπότε υπάρχουν διαφορές, κατά το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος διακριτικής μεταχείρισης, δηλαδή σε μια ξένη χώρα μπορεί κάποιος να έχει λιγότερη αποζημίωση. Τώρα, για τις διαταγές προστασίας, εντολές προστασίας των θυμάτων, έχουμε και εδώ πέρα κάποια μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης, κανονισμό των Ευρωπαϊκών Μέσων ε, Προστασίας ε, και την σχετική οδηγία, αλλά και πάλι τα μέσα αυτά δεν χρησιμοποιούνται πολύ και ε, δεν έχουμε τώρα τον χρόνο να τις δούμε αυτές τις εντολές, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορείτε να διαβάσετε. Κατόπιν, ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε από όλα αυτά. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουν αυτές τις διαφορές. Κάποια από αυτά δείχνουν ε, τύφλη εμπιστοσύνη, θα λέγαμε. Δηλαδή, θέλουν διασυνοριακή συνεργασία με οποιοδήποτε κόστος παραδείγματος χάνει όσον αφορά το παραδεκτό των τεκμηρίων δεν τους απασχολεί κάποια άλλα έχουν ε, μια προσέγγιση θα λέγαμε μεσοβέζικη καθώς ε, γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις αλλά θεωρούν ότι διαφυλάσσουν τα βασικά δικαιώματα. Και τέλος υπάρχουν κατημέλη τα οποία δείχνουν πλέον μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα και αυτό αφορά ιδιαίτερω τι ε, συνθήκες κράτησης. Πλέον κρατημέλη δεν ανέχονται παραβιάσεις του άρθρου 4 της ε, χάρτας. Ε, τι έκανε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπάθησε να υπάρξει μια σύγκληση όσον αφορά το δικονομικό δίκαιο Επίσης ε, έκανε κάποιες προσαρμογές, διεύρυνε το πεδίο εφαρμογή των μέσων συνεργασίας για να περιλάβει και τις διοικητικές αρχές και όταν δεν γινόταν αυτό απλά παρέπεμψε στο εθνικό δίκαιο αυτό παραδείγματος χάρη ισχύ όσον αφορά τη δυνατότητα νομικής προσφυγής η οποία δεν εναρμονίζεται. Οπότε, τι γίνεται. Είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα. όχι ιδιαίτερος. Εδώ πέρα βλέπετε μια σύνοψη των ζητημάτων που αντιμετωπίσαμε, παραδείγματος χάρη είχαμε μακροσκελείς διαπραγματεύσεις τέσσερα χρόνια για, τους, για την οδηγία και τον κανονισμό και είχαμε πολύ δραστικές περάκοπες όσον αφορά τα αρχικά μέτρα ερεύνης. Επίσης υπήρχε κακή εκτέλεση των ετοιμάτων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, δεν υπήρχε αμοιβαία γνώση, επικοινωνία ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι το οποίο τελικά κατέληξε σε κάποιες ασυμβατότητες μεταξύ των κρατών μελών και τέλος έχουμε τη μη αναγνώριση, τη μη χρήση των μέσων. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ε, πολλά από τα οποία έχουν μπλοκαριστεί. Ε, Αυτό ισχύει και για το, το Ευρωπαϊκό την οδηγία για την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας ε, αλλά και τα θέματα της προφυλάκησης όπου δεν υπάρχει κάποια μεγάλη επιτυχία. Αν θέλετε, λέει ο περάστε στις συστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ μεγάλη η έρευνα και έχουμε δύο εισηγητές ε, που οπωσδήποτε θα θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Όχι εντάξει, μην σταματάτε εντελώς. Απλά πείτε μας τα σημαντικότερα για να περάσουμε σε ερωτήσεις. Όσον αφορά τις συστάσεις, ε, προτείναμε έναν συνδυασμό φαινός ε, ήπιων μη νομοθετικών μέτρων και πρακτικών εργαλείων. Για τα πρακτικά μέσα, το σκεπτικό ήταν να υπάρξει κάποια εκπαίδευση και ενημέρωση και κυρίως ε, να απευθυνθεί αυτή η εκπαίδευση σε περισσότερους, να περιληφθούν δηλαδή και οι πάροχοι των υπηρεσιών, γιατί θα έχουν μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της συνεργασίας, όπως έχει δείξει η υπηρεσία για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια. Επίσης, ε, προτείναμε να εστιάσουμε σε κάποια από τα ευρωπαϊκά αυτά εργαλεία τα οποία δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα κάποια δημοσιότητα. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να περιληφθούν κάποια εργαλεία στήριξης και κάποια κατεύθυνση για όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά στην πράξη και βεβαίως διάλογο μεταξύ των δικαστικών αρχών οριζοντίου αλλά και κάθετο διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Επίσης επιμείναμε στο να αναπτύξουμε κοινοτική οικονομική στήριξη σε διάφορα μέσα, όπως ε, τα μέτρα ερεύνης, τις συνθήκες κράτησης, τους μηχανισμούς αποζημίωσης ε, για κράτηση και για τα θύματα διασυνοριακών υποθέσεων. Συνοψίζοντας τώρα όσον αφορά τις ε, νομοθετικές μας προτάσεις, επιμένουμε πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κωδικοποίηση του κεκτημένου, να δούμε τα και να εφαρμογής που υπάρχουν στο διοικητικό δίκαιο και μετά βρήκαμε πέντε τομείς όπου θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία βραχυπρόθεσμα. Πρώτα απ' όλα στο θέμα των συνθήκων κράτησης, να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες συνθήκες. Επίσης, ε, στο θέμα της παραδεκτότητας των τεκμηρίων, η ενίσχυση του πλαισίου για την ε, επανεξετασία από τα δικαστήρια όσον αφορά και την προφυλάκηση και το παραδεκτό των τεκμηρίων και βεβαίως ε, το θέμα της αποζημίωσης των συστημάτων αποσμίωσης για τα θύματα και για την αδικαιολογητή ε, κράτηση. Αυτά πρόθεσμα. Επίσης, ε, έχουμε και κάποιες πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ε, προτάσεις, αλλά εδώ θα σας παραπέμψω στην μελέτη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τι δύο. Θα έχουμε τώρα έναν λίγο χρόνο για ερωτήσεις. ήταν ε, η Κατερίνα Εκινίτση είναι η συγγήτρια, είναι μάλλον επικεφαλής ε, για τα ε, διαδικαστικά δικαιώματα για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντική η, η, εργασία που έχετε κάνει και το παράρτημα που έχετε προσθέσει με τις ε, ε συγκριτικές εκθέσεις για τις χώρες και πιστεύω πως θα βοηθήσει την, τους συναδέλφους που μελετούν το, το, το δικαιονομικό ε, ε, δίκαιο. Φαίνεται να είναι παράπλευρο θέμα, αλλά για τη δική μας Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό, μαζί και με όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Διάβαζα το κείμενο την ώρα που μιλούσατε ε, ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμο λοιπόν και έχω και εγώ μια ερώτηση. Εδώ είναι ε, δύο μέλη που θέλουν να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Η Μπρικίτ και μετά η Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ λεπτομερή μελέτη που μας βοηθά θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι ορισμένε φορέ έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αν η μελέτη είναι πολύ βοηθητική και μα δίνει πολλέ πληροφορίε, ίσω είναι απαραίτητο επίση να γίνει ένα είδος δημόσιας ε, εκστρατείας ε, μέσω των ε, ψηφιακών υπηρεσιών έτσι ώστε να μην τη γνωρίζουν μόνο οι ειδικοί στο Κοινοβούλιο αλλά να το γνωρίζουν περισσότεροι. Να διαδοθούν περισσότερο δηλαδή τα πορίσματα. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Είμαι ευτυχής που επίσης αναφέρατε στην εισήγησή σας την έκφραση της τυφλής εμπιστοσύνης, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο για εμπιστοσύνη, αλλά το θέμα δεν είναι η εμπιστοσύνη, αλλά είναι η ελλειπής γνώση των διαφόρων συστημάτων όσον αφορά τους ε, αναφέρονται και πολύ διαφορετικά νομικά και δικαστικά συστήματα. Εδώ το λόγο κάνουμε συζήτηση για την ε, ε, κράτηση την, πριν από την δίκη. Ε, έχουμε πολύ διαφορετικά συστήματα και γι' αυτά ε, θα πρέπει να συζητήσουμε. Και επίση έχω μια ερώτηση για τις αποζημιώσεις, γιατί η αποζημίωση είναι φυσικά ένα σημαντικό μέσο. Αλλά εάν κανείς έχει προφυλακιστεί σε πολύ πρώιμο στάδιο, ίσως να μείνει υποκράτηση και για ένα χρόνο. Και μετά με στέλνουν σπίτι μου όπου δεν ξεκινά καν κάποια διαδικασία εναντίον μου, αλλά ολόκληρη η ζωή μου έχει καταστραφεί. Τι είδου αποζημίωση λοιπόν μπορεί κανείς να προβλέψει σε τέτοια περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μία βήμα το βήμα προσέγγιση ώστε να αλλάξουμε το σύστημα σε κάποια από τα κράτη-μέλη γιατί αποζημίωση σημαίνει χρήματα. Αλλά δεν αρκεί, δεν αρκούν τα χρήματα. Συμφωνώ ότι χρειάζεται στήριξη για τα θύματα. Μιλήσατε για την προστασία των θυμάτων. Όμως νομίζω πως μετά από ένα έγκλημα θα πρέπει να σκεφτούμε, να σκεφτούμε τα θύματα γιατί συχνά βοηθάμε το δράστη να ξεπεράσει το, τα προβλήματά του αλλά όχι το θύμα. Και είναι αυτό πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τρομοκρατία αλλά και για όλα, όλα τα είδη βίας. Εδώ συμμερίζομαι τη γνώμη σας για τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, τη συνεργασία για να δούμε αν θα πρέπει να ζητήσουμε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή όχι, γιατί το νομικό σύστημα στην άλλη χώρα είναι τελείως διαφορετικό και Ω προ αυτό, μια τελευταία παρατήρηση, γιατί ο πρόεδρο ανέφερε τι αποδείξει. Συχνά είναι καλύτερο να επενδύσουμε σε ανθρώπου, σε γνώσει, σε περισσότερε δυνατότητε για τα συστήματά μα και έτσι βήμα το βήμα να τα εναρμονίσουμε τα συστήματά μα και όχι να βάλουμε και πάλι και πάλι νέα μέτρα όπω το Ευρωπαϊκό Ένταλμα το ε, έρευνα, συγγνώμη, όπου το έχουμε εδώ και ένα χρόνο μόνο, αλλά ξέρουμε ότι στην πράξη μπορεί να μην λειτουργήσει λόγω των διαφορών στα συστήματά μα λοιπόν τις προτάσεις σας και όπως είπα και εξ αρχής ίσως χρειάζεται επιπλέον ε, εκστρατεία ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ε, συνειδητοποίηση για αυτά τα θέματα. Πριν φτάσουμε στις αποδείξεις, ναι, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το ανθρώπινο στοιχείο που πολλαπλασιάζεται. Εγώ έχω κάποια ερωτήσεις για το EAW. Κατερίνα όμως πρώτα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, τις ε, προσκεκλημένες μας για την παρουσίαση αυτού της μελέτης. Πολύ ενδιαφέρουσα, ήθελα θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνος για να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Όμως θα συζητήσουμε για αυτά που ήδη μας είπατε, που είναι ήδη ε, πολύ σημαντικά. Για μας που δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα θέματα, να σας πω ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και έτσι όλες οι διατάξεις, όπως ας πούμε αυτά που ε, ανέφερε πριν η Birgit που προηγήθηκε, να μπορούν να ε, ισχύουν σε όλες τις χώρες. Γιατί διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν αποτελούν εμπόδιο. Εγώ θέλω να σας πω κάποιες και προβληματισμούς και να διαρωτήσεις. Ε, πιστεύω πως είναι σωστό αυτό που είπε η Μπίργκη ότι δηλαδή να γνωρίζουμε τα πορίσματα τέτοιων μελετών όπως αυτή. Δηλαδή, όχι μόνο μεταξύ εμπειρογνωμόνων, μπορεί να είναι χρήσιμο, όμως πιστεύω και είμαι βαθιά πεπισμένη, πως το είπαν και, και εσείς, ότι μια από τις σημαντικές πτυχές για να δημιουργηθεί ε, ε, μια δυνατότητα ευρεία ε, συνεργασίας και ε, δημιουργία ίσων όρων για τις ποινικέ διατάξεις σε όλα τα κράτη είναι η κατάρτιση. Η κατάρτιση είναι το πιο σημαντικό εργαλείο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη νομίζω. Τούτο λεχθέντος έχω δύο ερωτήσει: Μία λίγο πιο τεχνική φύσης και η άλλη γενικότερη. Η Πιο ε, συγκεκριμένη ερώτηση αφορά το σύστημα αποδοχής των αποδείξεων και των αποδεικτικών στοιχείων και θα ήθελα να γνωρίζω πώς πιστεύετε ότι διάφορες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη σε σχέση με τους κανόνες αποδοχής των ε, αποδεικτικών στοιχείων και εδώ μιλάμε ε, σε μορφές κανόνων αποκλεισμού ή μη αποδοχής των αποδείξεων πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις ε, διακρατικές έρευνες της μελλοντική Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εσείς ε, κάνατε σε αυτό το νέο οργανισμό που θα ενταχθεί εδώ σε αυτό το πλαίσιο. Ε, και θα επανέλθω στο θέμα των ανηλίκων. Θα ήθελα να επανέλθω και στο θέμα των ανηλίκων, αλλά εν πάση περιπτώσει για να είμαι σύντομη δεν θα το κάνω, αλλά να σταθώ στα δικαιώματα των θυμάτων. Και ως προς αυτό, εγώ συμμετέχω στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία και δουλεύουμε για την τελική μας έκθεση και ανάμεσα στα μέτρα τα οποία έχουμε σκεφτεί υπεριλαμβάνεται και αυτό της δημιουργίας ενός κέντρου συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακριβώς για να εγγυηθούμε ότι όλα τα θύματα ε, τρομοκρατικών επιθέσεων που μπορεί να είναι διαφορετικής εθνικότητας όπως είδαμε να μπορούν να έχουν το ίδιο είδος ε, ε, αποκατάστασης, αποζημίωσης σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. Ακόμα και την έχουν δεχτεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα προέλευσής τους. Ευχαριστώ Κατερίνα να θέσω και εγώ μια ερώτηση. Ε, όταν κάνετε μια τέτοια μελέτη, το θέμα κλειδί της αμοιβαία αναγνώρισης, και τα διάφορα μέσα, πώς αυτά οριμάζουν, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. κάποια στιγμή οριμάζουν αυτά τα μέσα. Στην αρχή, ας πούμε, είχαμε προβλήματα με την αναλογικότητα για τα μικρά δικήματα και ούτω καθεξής. Είναι όμως τόσο ένα σημαντικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό έγινε εδώ Στη συνέχεια είδαμε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης αρχίζει να γίνεται σεβαστό λόγω της κατάρτισης των δικαστών, των σωστότερων αποφάσεων και γενικότερα γίνεται σεβαστό και εν γέννη φαίνεται να είναι ένα από τα καλύτερα οικονομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Πώς βλέπετε να γίνεται αυτό σε άλλους τομείς και αυτό έρχεται και συνδέεται και με τα αυτά που είπε να δημοσιοποιηθεί περισσότερο πώς η εναρμόνιση βοηθά στην ομαλότερη λειτουργία και συνεργασία. Εσείς ας πούμε για τη δίωξη δικημάτων του αστικού κώδικα ε, πώς θα γίνει αυτό και έπειτα μιλήσατε για συνθήκες κράτησης. Υπάρχει τελικά ένας μεγάλος εξωτερικός παράδειγμα, ας πούμε, αν δούμε στη Γερμανία. αν εγώ ήμουν ένα γερμανικό δικαστήριο, όπου οι συνθήκες κράτησης είναι καλύτερες, ας πούμε, από τις άλλες χώρες, μπορεί εκεί να υπάρχουν περισσότερες καθυστερήσεις ή απροθυμία ε, ε, ε, να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης λόγω αυτού. Ή μήπως εάν βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης ολόκληρη την Ευρώπη και δημοσιοποιήσουμε ότι αυτή είναι η μεταχείριση που θέλουμε, δηλαδή να μην κατηγορείται το ίδιο το εργαλείο, να έχουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση κατάρτισης, συνθήκες κράτησης, είναι δηλαδή όλα αυτά τμήματα μιας μεγάλης εικόνας και να μην ε, ακολουθούμε αυτή τη δικασία που, που δέχεται επιθέσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύρρηψης και έχει ε, ε, μετατραπεί στο αποπέδι όλων των ε, ευρωσκεπτικιστών χωρίς λόγο. Μήπως δηλαδή θα πρέπει να, τα θέματα εναρμόνισης είναι πολύ βασικά έχουν να κάνουν με προδιαγραφές σε κάθε χώρα. Αλλά στην ουσία πρόκειται για θέματα σωστής εναρμόνισης που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη λειτουργεί πολύ καλά. Η εναλλακτική δε είναι πολύ άσχημη. Το να επανέλθουμε δηλαδή στη, σύμβαση του 57, όπου πολλοί κακοί άνθρωποι εγκληματίες ε, πέρασαν χρόνια μέχρι να συλληφθούν. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η Birgit Σίπολ. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μια μεγάλη ε, εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να δείξουμε πως το τελικά η εναρμόνιση των ε, συστημάτων έχει επιφέρει μεγάλο ωφέλη. λύνουμε τα προβλήματα, αλλά σας λέω ότι για τους πολιτικούς ήταν ε, μια ένα μεγάλο πεδίο ε, για ε, θυματοποίηση ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Και πάλι αν δούμε στην Γερμανία όπου υπάρχει συνταγματική διάταξη όπου δεν μπορείς να απελάσεις ας πούμε προς χώρες τον ύποπτό σου. Το ίδιο μάλλον συσχύει στη Σλοβακία Η ιδέα είναι ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενημερωτική εκστρατεία για τα μέτρα τα οποία υιοθετούμε μέσα στο πλαίσιο της ποινική διαδικασίας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο πλός πολίτης καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται όταν προσπαθούμε να εναρμονίσουμε και μιλάμε για αμοιβαία αναγνώριση. Οι συνθήκες κράτησης είναι μάλλον ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και το λέω αυτό γιατί διαρκώς στην Europol γίνεται λόγος για αυτές τις καθυστερήσεις, γιατί οι συνθήκες κράτησης. Και επανέρχεται αυτό το θέμα συνέχεια. Με ενδιαφέρει λοιπόν αυτό και το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Όταν έκανε την έκθεσή της η κυρία Κινίτσι, το ίδιο ισχύει. Θέλεις να να φυλακίσεις παιδιά. Όχι, πουθενά δεν θε να το κάνει αυτό βέβαια, αλλά ειδικά σε κάποιε χώρε ακόμη λιγότερο. Και έχουμε αυτή την εντύπωση ότι πρέπει ε, κάπως λοιπόν να σπρώξουμε εδώ, να το διαδώσουμε και θα είναι ε, μια επιτυχία της Ένωσης. Ε, ε να το με αυτο αυτό. Ξέρω, είμαι λίγο πολύ ενθουσιώδης πρωί-πρωί, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε σε αμυντική θέση. είναι ένα τομέα κυριαρχία, αλλά πρέπει να μοιραστούμε την κυριαρχία και να τα καταφέρουμε. κυρία Κινίτσι μίλησε για δικαστές. Οι δικαστές θέλουν να καταρτιστούν, θέλουν να καταρτιστούν και να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εμένα με λυπεί όταν έγινε η επίθεση κατά του ευρωπαϊκού εντάλματο σύλληψη. και το αναθεωρήσαμε και μετά κοιτάξτε τι έγινε. Είναι ο Χρυσό Κανόνα για ολόκληρο τον κόσμο. Just like the European arrest warrant, but you know. Um, so thank you very much. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλα. Για τις δικές παρατηρήσεις, κυρία. <clears throat> Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, καταρχήν, ε, για λανθασμένη αδικαιολόγητη κράτηση στις διασυνοριακές υποθέσεις. Έχουμε επιμείνει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά ποτέ δεν συζητήθηκε στην πραγματικότητα. Το EGTN, το EGN, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, έχει κάνει μια μελέτη που εντοπίζει τις βασικές διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Και κενά στις ε, διασυνοριακές ε, διαδικασίες. Εντοπίζει περιπτώσεις όπου ύποπτοι δεν έλαβαν αποζημίωση παρόλο ότι κρατήθηκαν αδικαιολόγητα κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων ή περιπτώσεις στις οποίες ήταν πολύ δύσκολο να λάβουν αποζημίωση από το εκτελών ή από το ετών κράτος μέλος. Μπορεί να μην έχουμε χρόνο σήμερα να πούμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, αλλά χρειάζεται να το προσέξουμε αυτό το ζήτημα. χρειάζεται κάποια συνοδευτικά μέτρα για να ε, ενταθεί, να τονιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα διασυνοριακά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, επιμόρφωση των δικαστών, δεν είναι μόνο οι δικαστές βέβαια. Υπάρχουν και οι δικηγόροι υπεράσπισης, για παράδειγμα χρειάζεται και αυτοί να ενημερωθούν καλύτερα, να εκπαιδευτούν καλύτερα. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν λίγες πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθεί η υπεράσπιση και να εκπαιδευτούν οι δικηγόροι. Συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών για τις δικονομικές εγγύησεις, περισσότεροι δικηγόροι δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Παρόλο ότι θα τους έδιναν σοβαρά επιχειρήματα αν τις γνώριζαν. Τώρα να επανέλθω στις δικές σας παρατηρήσεις και εσάς και τις δικές σας κυρία μου. συμφωνώ μαζί σας ότι η αμοιβαία αναγνώριση έχει οριμάσει κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν κάποια κείμενα, τα, κάποια νομιστικά κείμενα, τα οποία ε, ήταν πολύ επιτυχημένα, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Κάποιες αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί ρυθμίστηκαν. Για παράδειγμα, η αναλογικότητα, την οποία αναφέρατε εσείς, Πρόεδρε. Άλλες αδυναμίες δεν έχουν θεραπευθεί. Για παράδειγμα, οι συνθήκε κράτησης. Και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας βέβαια. Είναι θέμα λήψης πρακτικών μέτρων και εφαρμογή υφιστάμενων προτύπων από που όμω που έχουν προβλεφθεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από διάφορες επιτροπές αρμόδιες στην Ευρώπη. Πρέπει να λυθεί το θέμα των συνθηκών κράτηση μέσω ελάχιστων προδιαγραφών. Και πιστεύω ότι από αυτή την πλευρά πρέπει να αναλυθεί νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια για παράδειγμα, τη νομική βάση. Υπάρχει νομική βάση στη συνθήκη για να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον τομέα. Είναι ένα ερώτημα. Εμείς δώσαμε κάποια επιχειρήματα για να υπερασπιστούμε την ύπαρξη νομική βάση αυτό το θέμα στην έκθεσή μας. Η ΕΛΟΝΤΗ. για τις συνθήκες κράτησης και τις ελάχιστες προδιαγραφές υπάρχουν. Υπάρχουν τα προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απλά δεν εφαρμόζονται το πιο βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητα, πολιτικής βούλησης από πλευράς των κρατών μελών. Και σίγουρα χρειάζεται οικονομική στήριξη των κρατών μελών γιατί δεν θα επενδύσουν σε αυτό. Τώρα, για το θέμα του αποδεκτού των τεκμηρίων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην αρχική πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπήρχε ένας κανόνας παραδεκτού για μη παραδεκτού βασικά, για τεκμήρια τα οποία έχουν συλλεχθεί παρανόμως, αλλά διαγράφηκε στις διαπραγματεύσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει το πώς έχουν συλλεχθεί τα τεκμήρια. το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αμοιβαίας γνώσης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι, οι δικαστικές αρχές κάνουν ερωτήματα, διασυνορικά ερωτήματα, διότι δεν υπάρχει, ε, μάλλον έχει υποσκαθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά η αμοιβαία εμπιστοσύνη χρειάζεται για να πάρει απόφαση ένας δικαστής. Τελικά όλα καταλήγουν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην εμπιστοσύνη. Και όταν δεν υπάρχει αμοιβαία γνώση, θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουμε ελάχιστες προδιαγραφές. Είναι και αυτός ένας τρόπος ε, τα κράτη-μέλη να προβληματιστούν από κοινού για τις κοινέ διαδικασίες και τι αμοιβέ διαδικασίε. Ο πρόεδρο λέει ότι έχουμε πολύ λίγο πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μα. Οπότε ας τελειώσουμε. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω τις μαγικές λέξεις που αναφέρατε, την ε, ολιστική σφαιρική προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα τρόπο έχουν οριμάσει τα δικονομικά μέσα, θα μπορούσαμε να τα δούμε ως μια μαγική εργαλειοθήκη συνεργασίας την οποία έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό χρειάζεται να προωθήσουμε τις, την συμπληρωματικότητα μεταξύ των μηχανισμών αυτών. Αυτό ως νέο επόμενο βήμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δυο σας. Πολύ πλούσια και σημαντική αυτή η μελέτη είμαι σίγουρος ότι θα είναι χρήσιμη στις ε, εισηγητρίες μας για θέματα ποινικής δικονομίας. Ελπίζω ότι θα δοθεί περισσότερη σημασία σε αυτό το ζήτημα το οποίο ανταγωνίζεται στην προσοχή μας με πολλά άλλα θέματα. Ελπίζω πράγματι να καταφέρουμε να κάνουμε μαγικά. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να περάσουμε στο σημείο 16. Αργήσαμε λίγο, έχουμε πάρει μια μικρή καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη, πέμπτη είναι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ελνανάρς για να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης για το πρόγραμμα ψηφιακή Ευρώπη είναι ένα από τα τομεακά προγράμματα του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την καθυστέρηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η προηγούμενη συζήτηση. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε μια γνωμοδότηση για την έκθεση της ΣΥΤΡΕ για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη και εμείς πρέπει να δούμε ακριβώς τις πτυχέ αυτές οι οποίες αφορούν την Επιτροπή μας και το πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τι δυνατότητε της Ένωσης για τους υπερυπολογιστές, την τεχνητή νοημοσύνη και τις προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, κάτι το οποίο μας χρειάζεται και να υπάρχει επίσης ευρύτατη χρήση στην οικονομία και την ε, κοινωνία μας. Και τα αποφάσισαν αυτά οι υπουργοί στο Ταλίν Έχουμε ήδη το πλαίσιο της στρατηγικής της ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι ακριβώς να έχουμε τα μέσα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις σχετικές φιλοδοξίες. Και πρέπει να δράσουμε και να επενδύσουμε σήμερα γιατί η τεχνολογία και η ζήτηση της τεχνολογίας ε, όσον αφορά τους υπερυπολογιστές ε, προχωράει πολύ πιο γρήγορα από την ε, προσφορά. σε άλλα μέρη του κόσμου έχουν πολύ καλύτερες υποδομές. Εμείς έχουμε μια εξαιρετική κοινότητα τεχνητής νοημοσύνης. Και τέλος, ο κατακαιρματισμός και οι χαμηλές δημόσιες επενδύσεις κάνουν την οικονομία και την κοινωνία μας πλέον να κινδυνεύουν καθώς ε, είναι διασπαρμένες ε, αυτές οι εταιρείε. Και τέλος όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. και βεβαίω η βασική πρόταση την οποία θα ήθελα να εξετάσετε είναι ακριβώς η κυβερνοασφάλεια ε, να αποκτήσει ένα πιο σημαντικό ρόλο, κυρίως όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αναμένω βεβαίως τους ε, συναδέλφους ε, και ελπίζω να μας στηρίξετε για να έχουμε μια ισχυρή γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν Γερούν για τις δύο αυτές προτεραιότητες που ανέφερε ένα, μια συνάδελφο έχουμε που θέλει να μιλήσει και μετά θα ακούσουμε και την ε, Κομισιόν Μπίργκιτ και Τόμας. Σας ευχαριστώ. Μία-δύο γενικές ε, παρατηρήσεις. Έχουμε κάποιες ε, μικρότερες επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται, αλλά έχουμε μείνει λίγο πίσω και εγώ θα χαιρόμουν βεβαίως για να να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν λύσεις στην ψηφιοποίηση, σεβόμενοι πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, να μην αντιγράφουμε μόνο τα όσα υπάρχουν, αλλά να αναπτύξουμε και νέα στοιχεία. Επίσης υπογράμμισα το θέμα της ε, κυβερνοασφαλείας γιατί σε όλους μας αρέσουν τα εύκολα μπορούμε να ψωνίσουμε, να κλείσουμε ένα ξενοδοχείο, ένα ειστήριο από το σπίτι μας, όλα αυτά είναι ωραία και εύκολα, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι αυτός ο ψηφιακός κόσμος παράγει και νέες δυσκολίες όσον αφορά την ασφάλεια, την πρόσβαση στα δεδομένα, χειραγώγηση ανθρώπων και χειραγώγηση εκλογών. Και αν μπορούν να το κάνουν αυτό ένα-δύο μεγάλοι παίκτες ε, μόνοι τους ή να πουλήσουν τα δεδομένα, να χειραγωγούν δηλαδή ανθρώπους και εκλογές παγκοσμίω, αυτό σημαίνει ότι αν έχει κανείς λεφτά μπορεί να αγοράσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε έτσι ώστε τελικά όλοι μαζί, οι αρχές και οι πολίτες να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις νέες ε, δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα βεβαίως να μην ε, χειραγωγούμε, αλλά να προστατεύουμε και τα δικαιώματα των πολιτών μας. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα λεφτά βεβαίως προς την έρευνα και για να δώσουμε και την ευκαιρία στις μικρές επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα τέτοια στοιχεία. Εδώ πέρα μας έχουν βάλει πολύ σύντομη προθεσμία και νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, μας απασχολούν. Λοιπόν, θα πάει στην Ήτρια 16 Οκτωβρίου. Τόμας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω την ε, τσεχική βεβαίως. Ε, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαιτέρως ε, που μιλώ μετά την Birgit. Δεν αντιληφθήκα πλήρως ε, το εάν μιλάει για το πρόγραμμα αυτό της ε, νέας ψηφιακής Ευρώπης ή γενικά για κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούμε. Εάν μιλάει γενικά, συμφωνώ μαζί της. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα για το νέο αυτό πρόγραμμα. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω εμπλακεί σε κάποια ζητήματα τον έλεγχο των ευρωπαϊκών ε, δημοσίων οικονομικών. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που δεν είναι πολύ ε, αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να σκεφτούμε τον σκοπό του προγράμματος. Ε, συχνά λοιπόν βάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν εφαρμόζεται, ο κόσμος δεν ξέρει το πρόγραμμα ή τις όρους ή άλλες φορές οι όροι αλλάζουν οπότε θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί καλύτερα. Το άλλο σχόλιο είναι το εξής. Δεν θέλω εγώ να ρίξουμε χρήματα σε ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω το πρόγραμμα αυτό να βοηθήσει χώρες. Ο σκοπός είναι οι χώρες ε, να μπορούν να βελτιώσουν ε, την υποδομή τους. Πρέπει επίσης οι χώρες να φύγουν από το χαρτί να πάνε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. φορά δεν μπορούμε να στείλουμε έντυπα διαδικτυακά και χρειάζεται να πάει κανείς αυτοπροσώπος να υποβάλει έγγραφα σε ένα γραφείο. Λοιπόν, αν θέλετε να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να είναι αποτελεσματικό από την αρχή και θα πρέπει να έχει νόημα ευθύς ε, εξ αρχής ε, και σε ολόκληρη την περίοδο. Αυτό έχω να πω. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κύριος Μπρολιόλο. Η κυρία. Συγγνώμη. Ευχαριστώ προσεκτική ανάλυση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν και τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα εύστοχα. Θα πρέπει να στηρίξουμε το πρόγραμμα ιδιαίτερα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και την, την πτυχή της προστασίας των δεδομένων. Να πω επίσης και να καθησυχάσω τους τελευταίους ομιλητές για το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα δεν ξεκινά από το μηδέν. Ε, βασίζεται σε προγράμματα που ήδη υπάρχουν όπως το Σαφτελεκόμ που ενισχύει τον εξυγχρονισμό των ε, δημόσιων μηχανισμών και με το ΆΙΖΑ 2 εστιάζουμε επίση στους διοικητικούς μηχανισμούς. Θα βασιστούμε δηλαδή στα ήδη υπάρχονται και από εκεί ε, επεκτείνουμε και τη δράση τους. τα άλλα σχόλια που ακούσαμε και είδαμε μας βοηθούν στο να ενισχύσουμε το πρόγραμμα όσον αφορά το κομμάτι για την προστασία το... στο διαδίκτυο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα είμαστε σε θέση να λάβουμε υπόψη και να δεχτούμε τα περισσότερα σε σχόλια. Και εγώ το ελπίζω, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Φραντς μόλις ήρθε, θέλει να πει δύο λόγια και εκείνος και επανέρχομαι μετά στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη εκ πρώτη όψεω ε, μοιάζει φιλόδοξο 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ μοιάζουν πολλά αλλά σε βάθος 7 ε, ετών ε, κάθε χρόνο βγαίνει λιγότερο από το ετήσιο κέρδο της Google ή της Facebook. Τέλο πάντων, κάπου κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά θα πρέπει βεβαίω να είμαστε και λογικοί κάποια πράγματα για τις ε, παρατηρήσεις της ε, Λύπε. Η προστασία των ε, δεδομένων είναι πλέον νομοθετική υποχρέωση σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό. Και εδώ πέρα το άρθρο 6 θα πρέπει να συμπληρωθεί ή να υπάρξει και ένα ειδικό άρθρο. Δεύτερον, η κυβερνοασφάλεια θεωρείται από όλους ένα επιπρόσθετο εργαλείο. Δεν έχουμε όμως κατάλογα ε, εργαλεία για την ε, ασφάλεια τροφίμων. Είτε μιλάμε για τις ημερομηνίες λήξης είτε για τις αλυσίδες ε, ψήξης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σε όλους τους τομείς μια ανάλογη διασφάλιση, κάτι το οποίο απαιτεί και περαιτέρω κατάρτιση. Επίσης, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος ε, των ε, ψηφιακών ε, προϊόντων και να επενδυθεί ένα κομμάτι των χρημάτων στον έλεγχο του κώδικα πηγής του δωρεάν λογισμικού. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε να μην ενισχυθεί, να μην ενισχυθούν οι φυστάμενες διακρίσεις οι οποίες απλά θα περάσουν στους αλγορίθμους οι οποίοι μαθαίνουν μόνοι τους. Παραπέμπω εδώ πέρα στην έκθεση Big Data της κυρίας Κόμες. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να ολοκληρώσετε. Ναι, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Όταν εξετάζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, τα σχόλια ε, που ακούστηκαν από τους σοσιαλιστές και από τους πράσινους πιστεύω πως είναι κάτι που μπορούμε να προτείνουμε. Αν υπάρχουν λοιπόν προτάσεις για να ενισχύσουμε την γνωμοδότηση τις, ε, είναι ευπρόσδεκτες και επίσης σε σχέση με το οποίο ο Τόμας και ότι δηλαδή πρέπει να δούμε και την προστιθέμενη αξία ε, που θα ενισχυθεί από αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ωστόσο ότι χρειάζεται τις κυβερν... χρειάζονται οι κυβερνήσεις, οι δημόσιες αρχές και ο, δημο... και ο ιδιωτικός τομέας αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχει αυτό το πλαίσιο. Η, οι ΣΔΙΤ είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχία. Και σας ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω σε αυτό σε αυτή μας τη συνεργασία ώστε να πετύχουμε παρά το στενό χρονοδιάγραμμα. Ναι, το υπογραμμίζω κάθε φορά το στενό αυτό χρονοδιάγραμμα γιατί κάνουμε και το τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάθε φορά μας δίνουν ε, λίγο, λίγο χρόνο, ε, αλλά θα τα καταφέρεις, ε, Γερούν. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξετάζονται σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας. Ωραία, τώρα πάμε στην σε επιστροφές, ε, στην οδηγία για τις επιστροφές. Η Τζούτιθ είναι εδώ. Μόλις έλαβα την ενημερωμένη, τον ενημερωμένο κατάλογο σκιωδών. We move to the presentation now by the Commission of the proposal for. the... Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει την ε, αναδιατύπωση τη οδηγία για την επιστροφή των παραμών όμω διαμενόντων. Στι 12 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν υπέβαλε ένα ολόκληρο πακέτο προτάσεων που περιλαμβάνει και την ενίσχυση ε, της συνοριοφυλακής και ακτοφυλακή τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ανταπόκριση στις αποφάσεις του Συμβουλίου τη 28 Η Ιουνίου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σαρτζεντίνη. Πρώτα όμως θα ακούσουμε μια παρουσίαση από την Γενική Διεύθυνση Home, ο κ. Τιντεράτσι συγκεκριμένα θα μας κάνει μια παρουσίαση για ένα αριθμό θεμάτων συμπεριλαμβανομένων ε, γιατί δεν έγινε ε, του γιατί δεν έγινε μελέτη αντικτύπου για την αναδιατύπωση. Το εντοπίσαμε και το σχολιάσαμε παλιότερα. Θα μας μιλήσει και για άλλα θέματα βέβαια. Έχω και πολλέ απορίε, αλλά είμαι σίγουρο ότι η συγκήτριά μα θα τη στήξει από μόνη τη, δεν θα χρειαστεί να παρέμβω. Γενική κυρία Home, λοιπόν. Καταρχήν και μετά ο λόγος στην κυρία Σαρτζεντίνη. Χαίρομαι ότι ονομάστηκαν και όλοι οι σκιώδεις ηγητές πλέον, οπότε προχωράμε. Κύριε Τιντεράτσι, παρακαλώ. 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρίε και Είπατε ότι αυτή η πρόταση είναι τμήμα του πακέτου του Σεπτεμβρίου και έρχεται ως ανταπόκριση στα συμπεράσματα του, Ευρωπαϊκού, του Συμβουλίου του Ιουνίου. Επίσης αυτή η πρόταση κατά την άποψή μας είναι και η συνέχιση της, ε, που δίνουμε στην ε, εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Από το 2015 συγκεκριμένα έχουμε κάνει αποστολές ε, αξιολόγηση έγκεν για τα συστήματα επιστροφής στα 22 από τα κράτη-μέλη. Βασισμένοι σε τα πορίσματα αυτών των αποστολών, αυτών των επισκέψεων που ήταν τεχνικής φύσεως, αρχίσαμε να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα να, που δίνουν συνέχεια σε, σε, στην παλαιότερη δράση μας και θα πρέπει να μεταφραστούν σε νομοθεσία. Πέρσι για πρώτη φορά υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα που ήταν το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας, ένα βήμα προκειμένου να δώσουμε στα κράτη-μέλη πιο ήπια εργαλεία soft tools προκειμένου τα κράτη-μέλη να πιστούν να προσαρμόσουν τα συστήματα επιστροφής τους σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η σύσταση ακολουθήθηκε από πολλή δουλειά στην ομάδα επαφής με τα κράτη-μέλη για την τροποποίηση του εγχειριδίου ε, επιστροφών που ολοκληρώθηκε πέρσι το Σεπτέμβρη ενώ και αυτά ήταν όλα όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε σε επίπεδο ήπιων μέτρων. Τώρα, κοιτάζοντας τα πραγματικά νούμερα και την εξέλιξη των επιστροφών τα τελευταία χρόνια. Το συμπέρασμα φέτος ήταν ότι πρέπει να γίνει προσαρμογή και της ίδιας οδηγίας προκειμένου να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία και να ενταχθούν σε νομοθετικό πλέον κείμενο τα μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα σε εθνικό επίπεδο και δημιουργούν και τους κατάλληλους συνδέσμους ανάμεσα στο εθνικό επίπεδο και το κεντρικό επίπεδο τη Frontex για να αποκτήσουμε για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να σας αναφέρω τις επτά βασικές κατηγορίες αλλαγών που επιφέραμε στην οδηγία. Και μετά, αν θέλετε, δίνουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το α ή το β ζήτημα. Πρώτη κατηγορία αλλαγών έχει σχέση με τον δεσμό ανάμεσα στο άσυλο και τις διαδικασίες επιστροφής. Ενισχύουμε αυτό το δεσμό, αυτή τη σύνδεση. Έχουμε πλέον πιο αποτελεσματικούς κανόνες ε, για, το, για την ε, λήξη της ε, νόμιμης διαμονής ε, και την αφαίρεση της άδεια εργασία κλπ. Ε, κατόπιν μιας αρνητικής ε, απόφασης για το άσυλο, ε, πλέον συνδέουμε πολύ περισσότερο αυτή την απόφαση με την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής. Άμεση έναρξη της διαδικασίας επιστροφής συγκεκριμένα. Δεύτερη κατηγορία αλλαγών έχει σχέση με τα ένδικα μέτρα μέσα βασικούς, έχουμε σαφείς κανόνες πλέον ε, για ε, θέσεις, για προσφυγές ε, και εξετάζοντας την πρακτική και την ομολογία στα κράτη-μέλη διαπιστώνουμε μεγάλη διαφορά για το, στο, στο πώς η, τα, η χρήση ενδικών μέτρων και οι προσφυγές οργανώνται στα κράτη-μέλη και πλέον αποδίδουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου με αυτές τις αλλαγές. Τρίτη κατηγορία αλλαγών που σχετίζεται με μια καινούρια διάταξη για την υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών και πολιτών τρίτων χωρών. Ε, σε αυτό το άρθρο μάλιστα δίνουμε και ένα κατάλογο με τομείς στους οποίους αναμένεται αυτή η συνεργασία. Επίση, τα κράτη-μέλη, οι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών έχουν πλέον την υποχρέωση να δίνουν πληροφορίε σε υπηκόου τρίτων χωρών για το πώ θα γίνει αυτή η συνεργασία. Τι αναμένεται από αυτού του πολίτε τρίτων χωρών και ποιε θα είναι οι συνέπειε τη μη συμμόρφωση. Τέταρτη κατηγορία αλλαγών έχει σχέση με αλλαγέ που γίνονται στο σύστημα εθελοντικής αποχώρησης ενισχύουμε τους κανόνες για την περίοδο για την οποία μπορεί να γίνει αυτή. Έχουμε εξετάσει τα συστήματα των κρατών μελών πλέον και βλέπουμε ότι υπάρχει μια φαιά ζώνη ανάμεσα στους όρους με τους οποίους ε, χορηγείται αυτή η δυνατότητα και στους όρους με τους οποίους δεν χορηγείται. Εκεί θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε τις διάφορες. Επίσης υπάρχει πλέον υποχρέωση για δημιουργία συστήματος θελοντικής αποχώρησης, επιστροφή, συγγνώμη. Ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη ήδη είχαν τέτοια συστήματα, αλλά θεωρούσαμε ότι αν μπήκε ως νομική υποχρέωση από πλευράς τους θα ενισχυθεί αυτή η διαδικασία γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα προγράμματα εθελοντικής ε, επιστροφής θα πρέπει να είναι τα προτιμόμενα. Πέμπτη κατηγορία και πάλι εισάγουμε μια υποχρέωση, καινούργια υποχρέωση, για τα, τα κράτη-μέλη πρέπει πλέον να αναπτύξουν συστήματα που θα τους επιτρέψουν να επεξεργάζονται καλύτερα τις επιστροφές και επίσης θα τους επιτρέπουν να ενημερώνουν την Frontex, να δίνουν στοιχεία δηλαδή στη Frontex για να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο το έργο της. Στο ίδιο πακέτο άλλωστε γνωρίζετε ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Frontex στις διαδικασίες επιστροφής και πιστεύουμε ότι ε, η ανταλλαγή, η, η βελτίωση ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και, στην, και τη Frontex αποτελεί βασικό πυρήνα αυτή τη προσπάθεια. Έκτη κατηγορία αλλαγών έχει σχέση με την κράτηση. Ε, αναθεωρήσαμε τους κανόνες για την κράτηση με ένα ελάχιστο κατόφλι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δεν τροποποιήσαμε τα ανώτατα όρια, παραμένουν όσοι έχουν σήμερα, αλλά μειώσαμε το ελάχιστο κατόφλι στους τρεις μήνες. Γιατί, Γιατί κοιτάζοντας ε, τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανάγκη τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ε, διοργανώσουν την επιστροφή, την διαδικασία επανεισδοχής κλπ. Κάτι που δεν είναι εύκολο. Κοιτάμε τους, τις πρακτικές λοιπόν των κρατών και βλέπουμε ότι τρεις μήνες είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που χρειάζονται τα κρατημέλη για να διοργανώσουν την, να την επιστροφή. Μπορεί βέβαια αυτό να είναι μικρότερο αν ο, ο, ο της χώρας επιλέξει να αποχωρήσει εθελοντικά. Τελευταία κατηγορία αλλαγών ε, είναι μια καινούργια διαδικασία στα σύνορα, συνοριακή διαδικασία, η οποία θεωρούμε ότι συμπληρώνει τις συνοριακές διαδικασίες ασύλου που επίσης την χάνουν αναθεώρησης μέσω του κανονισμού διαδικασιών ασύλου. Το τελικό, η τελική μορφή των διαδικασιών για τις επιστροφές στα σύνορα θα συνδεθεί άμεσα στενά με τις καινούριες διαδικασίες παροχής ασύλου στα σύνορα. Θέλουμε να μην μείνει κανένα κενό ανάμεσα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου στα, άσυλο, ε, στα σύνορα και την έναρξη άμεση έναρξη της ε, διαδικασίας επιστροφής. Έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι κρατούνται, συλλαμβάνονται στα σύνορα να μπορούν να επιστρέφονται αμέσως μετά την απόρριψη του αιτήματο ε, ασύλου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου. Συγγνώμη. Σε ευχαριστώ. Περνάμε στην εισηγητριά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ αποφάσισα να ζητήσω αυτή την έκθεση γιατί θεωρώ ότι οι επιστροφές είναι τμήμα της διαδικασίας ασύλου εγώ το λέω αλλά εξαρτάται και το πώς το διατυπώνει κανείς και βλέπετε ότι δεν είμαστε επιτυχείς ε, όσον αφορά τις ε, επιστροφές ε, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό και όχι βεβαίω να επιστρέφουμε ανθρώπου σε χώρε στι οποίε δεν έχουμε ζήσει ποτέ. Λοιπόν, γιατί δεν είμαστε επιτυχεί, Γιατί η άλλη πλευρά δεν θέλει να δεχτεί του πολίτε τη και βεβαίω αυτό σχετίζεται με το ότι δεν υπάρχουν σε δίδυοι. Οπότε το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί εδώ πέρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε τις ε, δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις για τις ε, συμφωνίες επανεισδοχής, όπου τρίτες χώρες λένε να εντάξει να πάρουμε πίσω τους πολίτες μας, αλλά τότε να ανοίξετε κάποια νόμιμη ιδίωτα. Εγώ λοιπόν δεν θέλω μια οδηγία η οποία θα λέει ότι το πρόβλημα με τις επιστροφές είναι ότι δεν τους κρατούμε αρκετά. Λοιπόν, εκτιμώ το ότι υπάρχει ένα νέο άρθρο που λέει ότι πρέπει να υπάρξει διευκόλυνση των εθελοντικών επιστροφών και θεωρητικώς μπορεί να το έχουν πολλά κρατημέλη, αλλά στην πράξη ε, δεν υπάρχει. Το άρθρο σας εκεί είναι κάπως περιορισμένο, τα περισσότερα από τα άρθρα και ε, τις αλλαγές αφορούν το ότι το άτομο δεν συνεργάζεται με τις αρχές, ότι θα αναγκαστεί να επιστραφεί γρήγορα. Ένας ενδιαφέρον κατάλογος κριτηρίων για το πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάποιος είναι υποπτός φυγής και ένα από αυτά είναι έλλειψη οικονομικών πόρων ε, συγγνώμη δηλαδή. Ποιος ε, παράτυπος ε, μετανάστης ε, δεν έχει έλλειψη οικονομικών πόρων και ποιος από αυτούς δεν μπήκε παρανόμως. Δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς κάποια στιγμή κάνουν κάτι από αυτά που αναφέρει ο κατάλογος. Οπότε αυτό δεν μας βοηθάει εδώ. Αυτό το οποίο με βοηθάει είναι ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία της εθελοντικής επιστροφής. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να σταθούμε και κύριε Πρόεδρε η έκθεση αυτή α, την ανέλαβα πριν από λίγο καιρό μόλις οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει μια σωστή πολιτική επιστροφών ε, είναι κάτι για το οποίο δεν έχω κάποια αμφιβολία. Και τέλος κάτι άλλο. Ο αυτοματισμός που έχουν κάποια κράτη-μέλη, δηλαδή να υπάρχει μία απόφαση επιστροφής ε, με απαγόρευση εισόδου δεν είναι σωστό. Εδώ πέρα βεβαίως δεν υπάρχει σύνδεση αυτή, αλλά λέει ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί είναι πιο δύσκολο να φύγει κάποιος εθελοντικά, εάν μετά θα έχει απαγόρευση εισόδου. Υπάρχει λόγος για να φύγει κάποιος εθελοντικά, για να κάνει μια επανένωση οικογένειας μετά, παραδείγματος χάρη. Κάτι το οποίο μετά σημαίνει απαγόρευση εισόδου σε ολόκληρη την Σέγγεν για πολύ καιρό. Λοιπόν, αν θέλουμε να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν θέλουν να φύγουν και να διευκολύνουμε την αποχώρηση με τρόπο που θα είναι αποτελεσματικός. Ευχαριστώ. Um, uh, ευχαριστώ, Judith. Ναι, παρουσίασες ε, τις αρχές ε, αυτές και πρέπει να πω επίσης αυτό το οποίο είπες στην αρχή ότι ότι ανέλαβε αυτό το θέμα και πρέπει να γίνει σωστά βεβαίως. Βλέπω ότι έχουν οριστεί και οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ανέφερα στην αρχή. Η αξιολόγηση αντικτύπου. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Αλλά αν μπορεί να γίνει παράλληλα θα ήθελα να το σκεφτείς γιατί... Θα πρέπει να έχεις ε, και εσύ και οι σκιοδεσίγητες τα κατάλληλα μέσα για να προχωρήσετε το θέμα. Θέλω λοιπόν να καταγραφεί τώρα. Λοιπόν, σήμερα είπαμε να γίνει μια εισαγωγική συζήτηση και να ακούσουμε και την Κομισιόν. Αλλά έχουμε και τους κοιόδης εισηγητές, οπότε αν θέλουν να μιλήσουν Σίλβη και μετά η Δεν είναι σκιώδης εισηγήτρια, αλλά θέλει να μιλήσει. Να πείτε κάτι. Ναι. Είμαι σκιώδης για την ομάδα μου, ε, οπότε ε, ασχολούμαι το θέμα. Αυτή η οδηγία που έλαβε έτσι ε, ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς το 2018 ήταν ένα πολιτικό γεγονός, όχι μόνο δεν έχει μόνο τεχνικές ε, παραμέτρους. Να σας θυμίσω ποιο, ε, ποια ήταν, ποιος ήταν ο στόχος αυτής της οδηγίας. Η, η πτυχή την οποία θέλω να θίξω είναι ότι το ποσοστό, ο αριθμός των επιστροφών 36% δεν είναι στο επίπεδο στο οποίο επιθυμούσαμε, επιθυμούσε η οδηγία. Η δεύτερη πτυχή από την άλλη μεριά είναι να πούμε ότι αυτή η πολιτική επιστροφών, αν είναι αποτελεσματική, θα επιτρέψει να μειωθούν οι ροές. Θα εκφράσω τις αμφιβολίες μου για αυτό το στίχημα το οποίο βάζουμε. Δηλαδή ότι η καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας αυτομάτως θα έχει ε, ως αποτέλεσμα τη μείωση των αφήξεων. Δεν μου φαίνεται ότι είναι τόσο σίγουρο αυτό. Είναι υπομφισβήτηση. Κατά τη συζήτηση αυτών των 7 διαφορετικών τύπων αλλαγών που θα γίνει, ε, θα το ξαναδούμε. Η οδηγία πρέπει να είναι απλή στη χρήση της, να είναι συνεπής, λογικά. Αν θυμάστε, η Κομισιόν πριν από ένα χρόνο είχε δημοσίευσει ένα εγχειρίδιο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα την οδηγία. Προφανώς τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν, δεν άρκεσε αυτό το εγχειρίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα είναι πιο απλή, πώς θα σέβεται περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οδηγία Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ακριβής γίνεται για κάθε έναν από τους τομείς, επτά τομείς αλλαγών. Ευχαριστώ Σιλβί και ευχαριστούμε και για την υπενθύμηση του πώς λεγόταν η οδηγία. Ωραία, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος ζήτησε πάλι τον λόγο. Ορίστε. Ναι. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν. Έχω μία ερώτηση για το άρθρο 6. για τον κίνδυνο φυγής. Εκεί πέρα λέει ότι υπάρχουν τα εξής ε, κριτήρια. Ε, είναι ασαφές. Δηλαδή πρέπει να πληρούνται όλα αυτά τα κριτήρια. Ε, εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, αλλά θέλω κάποιες εξηγήσει από την Κομισιόν. Μετά, για την κράτηση, γίνεται μία αναφορά στο άρθρο 6. Άκουσα ότι η Κομισιόν έχει κάνει αξιολογήσει ε, σε, 22 κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ακούσω αν υπήρχαν ελλείψεις στα κέντρα κράτηση. Δηλαδή, αν δείτε τη Σουηδία, ακόμα και αν ανταποκριθούμε σε όλα τα κριτήρια του άρθρου 6, υπάρχει έλλειψη θέσεων κράτηση. Για ε, θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι απόψει. Ε, κύριε Λένα, θέλετε να μιλήσετε η συγγητριά μας ε, που η σκιώδης θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αναδιατύπωση, αλλά ε, έρχεται και λίγο αργά. είναι ένα, ένα καινούριο το φαινόμενο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό και ε, τώρα η πρόταση έρχεται λίγο αργά. Εγώ οπωσδήποτε έχω εμπιστοσύνη στον εισηγητή, αλλά γνωρίζοντας και τις δύσκολες διαπραγματεύσεις της αρχικής οδηγίας, δεν ξέρω πώς ε, θα τα καταφέρουμε. Μια χαμένη ευκαιρία λοιπόν. Ειδικά χτες να δούμε, είχαμε εδώ την ΕΑΖΟ, μας μίλησε για το ετήσιό της πρόγραμμα και τον Αύγουστο είχαμε ένα ποσοστό αναγνώριση 33% και ποσοστό επιστροφών 36%. Προβληματικό αυτό γιατί ε, ξέρετε τα μέσα των κρατών μελών δεν είναι άπειρα και απεριόριστα. Όλα τα χρήματα, όλες οι επενδύσεις ε, που πρέπει να γίνουν για ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν τις διαδικασίες αλλά μετά ε, δεν περιμένουν το αποτέλεσμα, τελικά αφαιρείται και περιορίζει έτσι τα διαθέσιμα κονδύλια για άτομα τα οποία αξίζουν προστασία. Οπότε συμφωνώ με την εισηγήτρια. Πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τις αποφάσεις να βοηθούνται. Και μπορούμε να το δούμε αυτό και στην αναθεώρηση, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ε, κάποια πράγματα και να είμαστε και ειλικρινεί ότι ε, έχουμε άτομα τα οποία δεν θέλουν να επιστρέψουν. Και βεβαίω ε, θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέφουν στη χώρα προέλευση. Ναι, ναι. Ήρθε αργά, ναι, είναι αναδιατύπωση, ναι, πραγματικά είναι πολύ οδυνηρό να επιστρέφουμε ανθρώπους. Ε, ε ναι, ε, όλα αυτά είναι προφανή. Αυτό είναι το σκληρότερο κομμάτι του πακέτου ασύλου, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Και να γίνει και αξιολόγηση αντικτύπου αλλά έχουμε μια εισηγήτρια η οποία θα ανταποκριθεί στην πρόκληση. Έτσι, Τζούντιθ, μπράβο. Γιατί ακριβώς έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και είναι δύσκολα, αλλά δικαίω λες ότι αυτό είναι από τα δυσκολότερα. Um, Εντάξει, ας το ξαναπούμε. Το προφανές είναι πολύ δύσκολο. Η ε, κυρία Γκυγιό μου υπενθύμησε τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Οπότε, Ποιος άλλος. Θα πεις και εσύ το προφανές, Μπριγκίτ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, ε, υπάρχουν δυσκολίες στην επιστροφή, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν με τέτοιες οδηγίες. Για παράδειγμα, δεν έχουμε συμφωνίες επανεισδοχής με όλες τις χώρες προέλευσης. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Μην οικοδομήσουμε μια οδηγία η οποία θα βαραίνει τα άτομα χωρίς να υφίστανται συμφωνίες με όλες τις χώρες προέλευσης. Αυτό είναι πολλές φορές το πρόβλημα και όχι το αν κάποιος επιθυμεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πολύ σωστά, είναι μία από τις δυσκολίες. Το είπε και η κυρία Σαρτζεντίνη. Αν θέλουμε να επιστρέφουμε άτομα, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν όλες αυτές οι δίωδοι, νόμιμες και μη. Επίση να σας πω και το εξής. Ο, ο, τίτλος λέει ότι είναι ε, συνεισφορά της Επιτροπής για τη συνάντηση των ηγετών στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Δεν αναφέρεται καθόλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτης. Οπότε στο συγκεκριμένο πολιτικό κλίμα ίσως αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Και επιστρέφουμε στην Κομισιόν, κύριε Τεντεράκη. Σημειώσαμε όλα τα σχόλια που έγιναν. Και θα τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια όταν συζητηθεί το κείμενο. Να σας πω όμως ποια είναι η άποψή μου για μερικά θέματα. Όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, οι επιστροφές είναι πάρα πολύ περιπλοκές, ένα πολύ περιπλοκό ζήτημα. Δεν πρόκειται η οδηγία αυτή να λύσει όλα τα προβλήματα. Ασφαλώς και πρέπει να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες και πολύ συχνά σα αναφέρουμε τις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Να μην ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να πιέζουμε προς πολλέ κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Τώρα για τα πολύ συγκεκριμένα θέματα που οποία σχολιάσατε. Δεν υπάρχει αυτοματισμός ανάμεσα στις επιστροφές και τις ε, απαγορεύσεις εισόδου. Δεν υπάρχει κανένας αυτόματος σύνδεσμος. Ε, ο κίνδυνος εξαφάνισης. Ένας, ένα από τα αντικειμενικά μας κριτήρια στο άρθρο 6 είναι και αυτός. Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί αυτός ο κίνδυνος μαζί με άλλα κριτήρια. Ο κατάλογος αυτός άλλωστε δεν είναι εξαντλητικός. Είναι κάποιες υποδείξεις προς τους δικαστές, συστάσεις παραγών, τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Αλλά ενδεχομένως ο δικαστής να έχει και τα δικά του κριτήρια. Στο δεύτερο τμήμα, μάλιστα του άρθρου 6, λέει, λέγεται ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση εξαφάνισης γίνεται κατά περίπτωση. Υπάρχει επίση μια σχέση του άρθρου 9 με το άρθρο 6. Περί κράτησης. Η, ο κίνδυνος εξαφάνισης επηρεάζει το αν θα διαταχθεί κράτηση. Αυτά τα δύο, το άρθρο 6 και το άρθρο 9, συνδέονται μεταξύ τους. Επίσης, έγινε μια ερώτηση για το κατά πόσον ως τμήμα της αξιολόγησης Σέγγεν που κάναμε, βρήκαμε προβλήματα σε ό,τι αφορά την χωρητικότητα του κέντρου κράτησης. Πέστο το Δεκέμβρη σας ενημερώσαμε, και κλεισμένο το θυρών να θυμάμαι καλά, για τα πορίσματα των ε, ε, της έρευνας που κάναμε. Οι εκθέσεις αυτές είναι απόρριτες, οπότε δεν μπορώ να αναφέρω χώρες, αλλά υπάρχουν θέματα μειωμένης χωρητικότητας στο κέντρο κράτησης. Ευχαριστώ πολύ, συγγήτρια. Υπάρχουν κάποια εκκρεμή θέματα τα οποία δεν έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου. Για παράδειγμα, πόσο, τι μπορεί να απαιτήσει κανείς από το άτομο το οποίο είναι προς επιστραφή, προκειμένου να βοηθήσει την επιστροφή του. Αν δείτε τα δικαιώματα των υπόπτων, δεν ζητάτε από ένα από, ε, υπόπτο μια ποινική υπόθεση να στηρίξει τις διαδικασίες με τρόπο που να βλάπτουν τα συμφέροντά του. Όμως, όταν μιλάμε για επιστροφές, υπάρχουν ένα-δύο πράγματα που η αναδιατύπωση προτείνει ή ε, υποδεικνύει ότι πρέπει να κάνουν οι ε, επιστρεφόμενοι. Θα δούμε αν αυτά, θα το σκεφτώ αν αυτά είναι αποδεκτά ή όχι. Δεύτερον, όταν συζητούμε για το ποινικό δίκαιο, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, προσπαθούμε να μην προτείνουμε ελάχιστες κυρώσεις προτείνουμε μέγιστες ή ελάχιστες μέγιστες, αλλά όχι ελάχιστες κυρώσεις. Ελάχιστη κράτηση για τρεις μήνες δεν νομίζω ότι είναι κάτι το υγιές, γιατί αντιβαίνει με τις αρχές που έχουμε ακολουθήσει σε άλλους φακέλους, θα το σκεφτούμε. Και μετά, οι επιστροφές είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως τα κράτη-μέλη δεν αφιερώνουν και πολύ χρόνο. πολλά κράτη-μέλη, επειδή έχουν ήδη πολύ αδήλωτη εργασία στη χώρα τους, δεν τους ενδιαφέρει να έχουν ένα ακόμα μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων διαμενόντων. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα επενδύσουμε σε κέντρα κράτησης και λοιπά. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Αλλά σίγουρα ένα, ένα από τα προβλήματα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να επενδύσουν. Ε, οι εθελοντικές επιστροφές είναι η λύση. Είδαμε με τις αρχές του Αμπιτζάν ότι δυσκολεύονται να δεχτούν πίσω ε, ε, άτομα τα οποία δεν επιστρέφουν με τη θέλησή τους γιατί δεν θέλουν να το πουν στην κοινή του νόμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι επιστροφές και πολύ δαπανηρές και ιδιαίτερα όταν κάποιος επιστρέφει με τρεις-τέσσερις φύλακε ή σωματοφύλακε μέσα σε μία πτήση χωρί να το θέλει. Ευχαριστώ πολύ καλή τύχη με τους, στη συναντήση με τους σκιώδει ηγητέ. να πω και κάτι άλλο. Προσπαθώ να διοργανώσω στο Στρασβούργο την ερχόμενη, α, συγγνώμη, την ερχόμενη εβδομάδα ή στο Στρασβούργο μια συνάντηση ε, σκιωδών εισηγητών, αλλά ακόμα δεν έχω σαφή εικόνα. Thank you. Do we have to suspend? Σας ευχαριστώ πολύ. We have the next point um, on the reuse of public sector information. Επόμενο σημείο είναι η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Ο κύριος Κοράου δεν είναι εδώ. Pause until... Παύση μέχρι τις 11 διάλειμμα. Γιατί ο εισηγητής μας δεν έχει φτάσει. Στις 11 τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.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 So, Συνάδελφοι, ας πάμε στο σημείο 18, την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Εμείς ε, γνωμοδοτούμε υπό το ε, άρθρο 53. Εισηγητής είναι ο κύριος Κοράου και θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση. Από πλευράς ε, της Επιτροπής έχουμε τον κύριο Βόλμαν που είναι παρόν και θα δώσω νομίζω το λόγο πρώτα στον κύριο Κοράου. Κάντε εσείς λοιπόν πρώτα την παρουσίαση και μετά θα πάμε στην Επιτροπή. Δεν θα κάνω εισήγηση τώρα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ κατευθείαν να κάνετε την εισηγήσή σας. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, όσο γίνεται πιο σύντομος. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας για την χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Συμφωνώ για την ανάγκη ενημέρωσης της οδηγίας του 13 για να διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογή ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι δημόσιοι τομείς και έτσι να διευκολυνθεί όσο γίνεται περισσότερο η χρήση των πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και να εναρμονιστούν οι όροι για να ε, διατίθενται αυτές οι πληροφορίες. Η ομάδα όμω στηρίζει την ε, αρχή της ελεύθερης πρόσβασης της πληροφορίας, όταν αυτό σημαίνει καλύτερη προστασία και υπηρεσία προς τους πολίτες ε, όταν χρησιμοποιούνται και την έρευνα και την ανάπτυξη, πάντοτε όμως λαμβάνοντας υπόψη ε, τους όρους ε, που ισχύουν για την παροχή αυτών των δεδομένων. Εδώ έχω ασχοληθεί με τα πτυχές που αφορούν την προστασία των ε, δεδομένων που που γίνονται πλέον δημόσιο κτήμα και συνεργάστηκα με τους αρμόδιους. Θέλησα να εξασφαλίσω ότι η πρόταση αυτή ε, αντικατοπτρίζει την ισορροπία ανάμεσα στην χρήση αυτών των πληροφοριών αλλά και στην προστασία των δεδομένων. Θέλησα επιπλέον να αποφύγω τον κίνδυνο από, ερμηνείων από όπως από αυτές που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε θέματα προστασίας δεδομένων, πάντοτε με στόχο τη σωστή εφαρμογή αυτής εδώ της πρότασης. Αναφέρομαι για παράδειγμα στους ορισμούς των προσωπικών δεδομένων ή των ανώνυμων δεδομένων. Αυτό αναφέρεται στο γενικό κανονισμό που άρχισε να ισχύει φέτος τον Μάιο. Τέλος, όσον αφορά τα αποκαλούμενα ευαίσθητα στοιχεία όπως ορίζονται από το άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα για τον υγειονομικό τομέα, ε, ζήτησαν να εισαχθεί και μια αξιολόγηση κινδύνου που θα πρέπει να κάνουν οι εταιρείε ή μάλλον οι οργανισμοί ε, που θα ενταχθούν σε αυτήν την οδηγία. Δηλαδή, ποιον αντίκτυπο θα έχει η δημοσίευση αυτών των στοιχείων, ώστε να προστατευτούν όσο γίνεται περισσότερο. Θέλουμε να σεβαστούμε και τις διατάξεις του γουκου που δηλαδή ε, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Ελπίζω πως, ε, ε, μάλλον να ευχαριστήσω τους κοιόδες που συνεργάστηκαν μαζί μου αγαστά ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Κορέο. Έπρεπε εξ να αναφέρω ε, τη φύση της πρότασης, την αναδιατύπωση δηλαδή, ε, είναι ε, σύμφωνα με το άρθρο 104 και 105 του κανονισμού. Τροπο, τροποποιείται ένα τμήμα της πρότασης και αναπερίπτωση. Και αυτό αν είναι απαραίτητο για πιεστικούς λόγους, λόγω της εσωτερικής συλλογικής των τροπολογιών. Ε, άρα λοιπόν αυτό οι λόγοι, η αιτιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύουν την ε, κάθε τροπολογία. Εξ του Έλεκος και Όδης είναι ο κύριος Μπέκερ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την αναμονή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Μάικλ Μπόνι που είναι ο σκιώδης του ΕΛΚΑ για αυτό το θέμα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησής του και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μας. Η οδηγία PSI είναι ένα βήμα μπροστά για την επέκταση της νέας χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου τομέα ως τμήμα της οικονομίας των ευρωπαϊκών δεδομένων. Ε, στόχος είναι να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί περισσότερη νέα χρήση ε, ε, ε, επέκταση κάποιων από το, των ε, ορισμένων διατάξεων της οδηγίας ώστε να καλύπτονται δεδομένα ερευνητικά και να ε, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν τα στοιχεία. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι διαδικασίες θα σέβονται τους κανόνες του, δίκαιο, του θεμητού ανταγωνισμού και οι, νέες, οι νέοι όροι θα εξασφαλίζουν και τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα συστήματα, τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα για νέα χρήση για... θα πρέπει ο δημόσιο τομέα να μπορεί να διαθέσει δυναμικά δεδομένα όσο γίνεται πιο σύντομα μέσω σύγχρονων interface API και να διευκρινίζει την ανάκριση του κόστους της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων σε ένα περιθωριακό κόστος για την χρήση των δεδομένων αλλά και την απόλυτη προστασία των δεδομένων. Ε, οι κανόνες περί νέας χρήσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν ε, να τηρούν πλήρως τα δικαιώματα για τον ιδιωτική ζω... της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των, προσωπικών δεδομένων σύμμορφα προς την Ευρωπαϊκή Σχετική Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέικερ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Ο κύριος Βόλμαν από την Επιτροπή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης και για την υποστήριξή του για την πρόταση. Η έκθεση εστιάζει στην προστασία των δεδομένων, δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία, ότι η οδηγία για τη νέα χρήση των στοιχείων από το δημόσιο, του τομέα θα πρέπει να γίνεται με βάση όμως την προστασία των δεδομένων. Δεν είναι αντίθετες έννοιες ε, πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είναι τμήμα μιας ε, συνειδητοποιημένης και ενεργητικής ε, μορφής χρήσης των δεδομένων από το δημόσιο τομέα. Θα ε, ήθελα επίσης να τονίσω τις θετικές πτυχές αυτής της πρότασης και τον αντίκτυπο που θα έχει όχι μόνο ως μέσο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης αλλά και για τις ΜΚΟ, για τους ίδιους πολίτες. Δηλαδή ανοιχτά δημόσια στοιχεία δεν θα σημαίνει μόνο νέες υπηρεσίες πληροφόρησης και ε, στοιχεία. Δεν θα οδηγήσει μόνο στην πρόθεση της ε, τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη αλλά θα σημάνει και περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στα ε, ε, δημόσια θέματα. Ευχαριστώ κύριε Σκοράο αν το επιθυμεί και πάλι. Ωραία λοιπόν. Ε, η προθεσμία είναι, για την υποβολή των υπολογιών είναι 18 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Now move to um, another Σημείο 19. Um, uh, Παρουσίαση από πλευρά τη Κομισιόν. Στι 31 Μαου η Κομισιόν πρότεινε ένα καινούριο κανονισμό για την ανταλλαγή, συνδρομή και κατάρτιση για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κυβδηλία για την περίοδο 2021-2027. Το επωνομαζόμενο πρόγραμμα Περικλής 4 βασίζεται στο άρθρο 133 της Συνθήκης που προβλέπει μια έναρξη 1η Ιανουαρίου 2021. Είναι η συνέχεια του προγράμματος Περικλής 2020 προκειμένου να προστατευθούν τα καρτονομίσματα και τα νομίσματα του ευρώ από την παραχαράξη και την κυβδηλία. Δεν έχει γίνει μελέτη αντικτύπου. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ σε σχέση με αυτό. Τα ευρώ σε σημερινές τιμές θα είναι ο προϋπολογισμός. Το παλιότερο πρόγραμμα ήταν 7.344.000 ευρώ. Δεύτερον, προτείνεται ε, η, εφαρμογή του, ε, του κανονισμού ε, και για τις μη συμμετέχουσες χώρες στο ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 352 της συνθήκης. Ο κύριος Ντε είναι εισηγητής και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί εγώ δεν έχω παρακολουθήσει πολύ το ζήτημα. Κύριε Ντε είστε εισηγητής και για τα, τους δύο φακέλους Θα σας δώσω το λόγο, αλλά πρώτα ας μιλήσει η Κομισιόν. Ο κ. Γιώργαν Κάου. από την Κομισιόν. Thank you. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα Περικλής 4. Η πρόταση αυτή εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, διότι υφίσταται ακόμα σημαντική απειλή παραχάραξης. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έκτους δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 300.000 ε, έχουν εντοπιστεί 300.000 παραχαραγμένα ε, χαρτονομίσματα. Το 2015 βέβαια ήταν 450.000, έχει μειωθεί ο αριθμός, με, βέβαια με, τις, με την σειρά χαρτονομισμάτων τα χαρακτηριστικά ε, ε ασφαλείας αυξήθηκαν, οπότε αυτό μπορεί να, μειώσει, να οδηγήσει και σε μείωση. Ε, χρειάζεται όμως και πρόληψη και αυτή η πρόληψη προβλέπεται μέσω του προγράμματος Περικλής 4 έτσι ώστε να μετριαστεί η απειλή. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την τέταρτη γενιά προγραμμάτων Περικλής. Μια ενδιάμεση αξιολόγηση έγινε για, την, για το πρόγραμμα του 2000 ε, μέσω ενός ε, ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και αυτή η αξιολόγηση έγινε, ε, ε, έδωσε ως αποτέλεσμα ότι το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει τη δράση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των διοκτικών αρχών μεταξύ αυτών και ταυτόχρονα αξιολογείται ως Ε, ως θετικό και, ο, και αναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα ότι οι δράσεις θα πρέπει να συνεχιστούν για να μην κινδυνεύσει το ευρώ. Τέλος, το πρόγραμμα αυτό λαμβάνει χώρα με συνεργασία ε, διοκτικών αρχών, κεντρικών τραπεζών, κέντρων ανάλυσης είτε των κεντρικών τραπεζών είτε άλλων ανάλυσης των παραχαρακτέντων ε, χαρτονομισμάτων και βέβαια ιδιωτικών φορέων. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα ευρείας συνεργασίας και μάλιστα πολυεπιστημονικής συνεργασίας. Οπότε συμπληρώνει το αμείο όπως το ΤΑΙΚΣ ή το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας η Κομισιόν στο έγγραφο εργασία προσωπικού που υποκατέστησε την μελέτη επιπτώσεων εξέτασε μια σειρά πτυχών τις οποίες συμπεριέλαβα εργότερα στο ανακοίνωση του 2017. Επίσης οργανώσαμε μια δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα Περικλής 4, κατά τη διάρκεια της οποίας λάβαμε 30 συνεισφορές, 30 γνώμες ιδιωτών, αλλά και κρατικών αρχών, οι οποίες επένεσαν την πρωτοβουλία συνέχισης του πρόγραμματος Περικλής 2020. Για τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, η νομική βάση είναι το άρθρο 133, όπως αναφέρατε πρόεδρε, με την συνήθη ε, διαδικασία ε, και με γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Γενικής Τράπεζας που έχει δισταλεί στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Δύο εθνικέ δράσεις έχουμε. Τα κράτη-μέλη είναι μαζί με τις διοκτικές τους αρχές στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της παραχάραξης, όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης του 1929, όλα τα συμμετέχοντα κράτη της Σύμβασης και, όλα τα, και τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν επικυρώσει, πρέπει να έχουν ένα εθνικό κεντρικό γραφείο για το συντονισμό των αστυνομικών ερευνών για θέματα παραχαράξεις νομίσματος προκειμένου να προστατευτούν τα νομίσματα, όλα τα νομίσματα, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ένα διεθνές νόμισμα και το ευρώ είναι διεθνές νόμισμα, το ενιαίο κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς χρειάζεται μια δράση και σε άλλο ένα επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν του εθνικού επίπεδου. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν ζητά να συνεχιστεί το πρόγραμμα Περικλής και μετά το 2020. Άλλωστε, συνάδει και με, το, με τη δράση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και με το ΤΑΙΑΞ. Τώρα, πώς έχει το πρόγραμμα, τι μορφή έχει. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποτελεί συνέχεια του Περικλής 2020 κανονισμού δηλαδή 331. Εστιάζεται στην προστασία τόσο των νομισμάτων όσο και των νομισμάτων του ευρώ. Πέρσι 170 περίπου χιλιάδες παραχαραγμένα νομίσματα εντοπίστηκαν, μιλώ για νομίσματα που κυκλοφορούν. Εντοπίστηκαν τόσα νομίσματα αλλά και πάρα πολλά νομίσματα και χαρτονομίσματα πριν ακόμα κυκλοφορήσουν. Μετά από αστυνομικέ εφόδους και κατασχέσεις. Η παραχάραξη επηρεάζει και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο όχι μόνο να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, αλλά να συνεργαστούμε και διεθνώς με άλλες χώρες. Η, επιμείναμε, για παράδειγμα, η αρμόδια κεντρική αρχή της Ισπανίας να συνεργαστεί με χώρες της Νότιας Αμερικής, διότι οι χώρες της Νότιας Αμερικής πρωτοστατούν σε παραχαράξεις τόσο του ευρώ όσο και του δολαρίου. Πολλές παράνομες οργανώσεις, κυρίως στην Κολομβία, που ξεπλένουν χρήμα και μεταξύ άλλων παραχαράσουν και νομίσματα. Χρειάζεται λοιπόν να στηρίξουμε τις εθνικές αρχές και στην Κολομβία και στο Περού για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο. Ιδιαίτερα προφανώς θα εστιάσουμε στην προστασία του ευρώ. Συνεργασία επίσης και με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, οι οποίες από την άλλη μεριά έχουν ως προτεραιότητα την προστασία του δολαρίου. Εμείς, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ και τις εθνικές αρχές κρατών όπω όπως η Γαλλία και η Ιταλία, προσπαθούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά το έργο αυτό σε συνεργασία με τις χώρες Λατινικής Αμερικής για την προστασία του ευρώ. Όπως σας είπα, πρόκειται για μια ευρεία συνεργασία πολλών κλάδων τόσο στο 20 στο Περικλής 2020 όσο και στο Περικλής 4 προτείνουμε. Πρώτη γραμμή μάχης είναι η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές. Μετά έχουμε τις Εθνικές Αρχές και τις Κεντρικές Τράπεζες, τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης, Νομισμάτων και Χαρτονομισμάτων και τέλος ερευνητικά κέντρα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούμε ένα κοινό πρόγραμμα του γερμανικού και του γαλλικού νομισματοκοπίου που έχει σχέση με την παραχάραξη των διμεταλλικών νομισμάτων τα οποία αποτελούν σύνηθες θύμα και προτιμούμενο θύμα των παραχαρακτών. Ε, ε, οι, οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι ίδιες με το προηγούμενο πρόγραμμα, ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μέσω σεμιναρίων για παράδειγμα. Τεχνική συνδρομή στις αρχές που χρειάζονται συνδρομή για την ανάλυση, για παράδειγμα, των νομισμάτων και των χαρτονομισμάτων που έχουν παραχαραχθεί. Επίση χρηματοδοτούμε και την έρευνα. Αυτές είναι επιλέξιμες δράσεις. Τέλος, έχουμε χρηματοδοτήσει και την αγορά εξοπλισμού. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης μπορούν να αγοράσουν εξοπλισμό προ χρήση μέχρι και τρίτων χωρών αν το επιθυμούν προκειμένου σε τρίτες χώρε να εντοπίζονται παραχαραχθέντα νομίσματα και χαρτονομίσματα. Η Ιταλία το έχει κάνει αυτό α πούμε, έχει αγοράσει εξοπλισμό με αυτή τη χρηματοδότηση ε, και αυτό ο εξοπλισμό χρησιμοποιείται από το Μοντενέγρο, ε, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο, παρόλο που δεν ανήκει προφανώ στη ζώνη του ευρώ, έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί το ευρώ και βοηθήθηκε από την Ιταλία σε θέματα εξοπλισμού. Τώρα για την εφαρμογή. Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται η ίδια η Κομισιόν. Ε, το ποσοστό συγχρηματοδότηση είναι 70% μέγιστο. Σε ειδικέ περιστάσεις μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 90% και οι επιχορηγήσεις είναι άτοκες. Επίσης, σε ό,τι αφορά θέματα προμηθειών, η Κομισιόν αυτό που έχει κάνει είναι να διοργανώσει ειδικές συνεδριάσεις με ενδιαφερόμενους ε, με ειδικευμένε εταιρείε ε, του κλάδου ε, προκειμένου να βελτιωθούν οι αισθητήρε εντοπισμού παραχάραξης των νομισμάτων. Οπότε βοηθούμε και τον κλάδο συγχρηματοδοτώντας ή χρηματοδοτώντας 100% σεμινάρια προκειμένου να ε, βελτιωθούν οι τεχνικές μας. Ετησίως υιοθετούμε ένα πρόγραμμα δράσης. Έχουμε και κάποια καινούργια στοιχεία στο καινούριο πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση για παράδειγμα. Έχουμε πλέον δείκτες απόδοσης, τρεις συνδεδεμένοι με ποσοτικά στοιχεία, ένας με ποιοτικό στοιχείο και μέσω κατεξιοδότηση πράξεων μπορούν ε, μάλιστα να ε, τροποποιηθούν, να ε, επικαιροποιηθούν αυτοί οι δείκτες από την Κομισιόν. Αυτά για την πρότασή μας. Αν μου επιτρέπει ο χρόνος... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάμε τώρα στον κύριο Ντεγιόγκ, τον εισηγητή και για τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γενικός στόχος ε, του προγράμματος αυτού νομίζω είναι κάτι το σημαντικό. Οπωσδήποτε η παρχάραξη του ευρώ είναι μια σοβαρή προτεραιότητα για όλους μας και για όλα τα κράτη-μέλη του του ξεκινήσατε λέγοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπήρχε αξιολόγηση αντικτύπου. Και πρέπει να πω ότι το να λαμβάνουμε ένα έγγραφο εργασίας ε, του προσωπικού δεν είναι το ίδιο με μια επίσημη αξιολόγηση αντικτύπου, την οποία θα ήθελα, γιατί όλες μου οι παρατηρήσεις αφορούν περισσότερο την ε, πτυχή του προπολογισμού. Αλλά βεβαίως ε, το θέμα είναι ακριβώς ε, το πώς θα έχουμε μια σωστή χρήση των κονδυλίων. Η πρώτη παρατηρήση που έχω να κάνω είναι ότι ο στόχος του προγράμματος η πρόληψη και η καταπολέμηση της παραχάραξης και της κινδυλίας, εντάξει. Αλλά μετά λέει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης καθώς ενισχύει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν διαφωνώ, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι για πολλούς που κοιτάνε το τι κάνουμε εμείς εδώ, γεγονό ότι έχουμε ένα πλαστό ευρώ για να τους πει ο καταστηματάρχης έχετε πλαστό νόμισμα. Αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου. Δηλαδή είναι θέμα που πάει πέρα από την ε, ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Είναι θέμα εμπιστοσύνη ε, στο χρήμα. Πρέπει να το διευρύνουμε λοιπόν κάπως. Τώρα για τον προϋπολογισμό την πλευρά ελέγχου του προπολογισμού. Κοίταξα το παράρτημα, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε δείκτες απόδοσης, ε, να έχουμε μια επιχειρηματική προσέγγιση. Και έχουμε κάτι το πολύ μικρό, μισή Το πρώτο είναι, λοιπόν, ο πρώτος δείκτης είναι αριθμός ανιχνευτέντων πλαστών ε, ευρώ. Αν ακούσω λοιπόν ότι υπάρχουν περισσότερα πλαστά ευρώ, τι σημαίνει, το πρόγραμμα είναι επιτυχές ή όχι. Γιατί όσο περισσότερα πιάνεις, τόσο περισσότερο έγκλημα υπάρχει. Οπότε τι κάνει το πρόγραμμα για να καταπολεμήσει αυτό το έγκλημα, γιατί και αυτό είναι το μέρος ε, του προγράμματος. Οπότε θεωρώ ότι οι δείκτες δεν μου λένε κάτι για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, αλλά για την κατάσταση όσον αφορά την πλαστογραφία. Και αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε εγώ θέλω να γνωρίζω υπάρχει κάποια απόδοση των χρημάτων μας. Ε, τώρα θα προσπαθήσω λοιπόν η έκθεσή μου να τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά, ε, να αποσαφηνίσει ότι υπάρχουν διαφορετικές πτυχές ε, που βεβαίως ε, πάνε μαζί. Δηλαδή υπάρχει πρόληψη, η προστιθέμενη αξία, να γνωρίζει ο κόσμος και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την κυβδηλία Και βεβαίω μετά υπάρχει και η επιβολή. Και όταν φτάνουμε στην επιβολή δεν είναι μόνο τα εθνικά κρατημέλη και η ΕΚΤΑ, αλλά έχουμε και τη Γύροπολη. Και είναι δύσκολο να αντιληφθώ. Εντάξει, πάντα αυτά είναι συμπληρωματικά, πάντα παραπέμπουν σε άλλους φορείς, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ πού ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα της επιβολής. Ε, και το τι ε, έχει κάνει η Europol. Ξέρω ότι κάνει αρκετή δουλειά. Και ακριβώς εδώ πέρα βλέπουμε ε, το ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την διπλή χρηματοδότηση γιατί υπάρχουν από διάφορες πηγές ε, ε, λεφτά τα οποία πηγαίνουν σε διάφορα προγράμματα. Μπορεί να υπάρχει διπλή χρηματοδότηση λοιπόν και δεν υπάρχουν κάποιες εγγύησεις. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Αυτά λοιπόν, στήριξη για το πρόγραμμα. Ε, δεν ήξερα ότι η Europol είχε τέτοιες ε, αρμοδιότητες. Ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τσινίτση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που σήμερα μας παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα το οποίο όπως ήδη υπόθηκε και από τον συνάδελφο εισηγητή είναι ένα πρόγραμμα σημαντικό βέβαια ε, γιατί Νομίζω πως η προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας σημαίνει όχι μόνο ότι δίνουμε και στους πολίτες βεβαιότητα σε σχέση με το νόμισμα που χρησιμοποιούμε, αλλά σημαίνει και την αναχέτηση της ε, διεθνούς, του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος που συχνά κάνει τέτοιου είδου ε, αδικήματα. Ο συνάδελφος ε, υπογράμμισε τις αντιρρήσεις ε, που έχει και παρατηρήσεις, ε, πράγματα για τα οποία και εγώ συμφωνώ. Ωστόσο, παραμένει ότι το πρόγραμμα, γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί δεν είχαμε κάνει ε, αξιολόγηση κινδύνου. Ίσως θα πρέπει λοιπόν εδώ να μας προβληματίσει αυτό. Ε, επίσης, συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις που σχετίζονται με τους δείκτες επιδόσεων. Ίσως αυτό το πρόγραμμα, αλλά είναι και περισσότερο, να ανταποκρίνεται στους στόχους για τους οποίους μιλήσαμε. Η Κομισιόν στην εισηγησή της αναφέρθηκε και την ύπαρξη μιας ολοένα και μεγαλύτερης εξωτερικής διάστασης των κέντρων ε, παραχάραξης, εξωτερικής εννοώ της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Πιστεύω πως ε, αυτή η αξιολόγηση λοιπόν ε, θα πρέπει να πάει όχι μόνο για την Λατινική Αμερική, αλλά και όπως έδειξαν πιο πρόσφατες έρευνες και προς τις χώρες της Μεσογείου, τα Βαλκάνια ή και την Κίνα, όπου πιο πρόσφατα ε, ε, αναγνωρίστηκε ως κέντρο παραχάραξης. Μια αναφορά ε, έγινε για την απέτηση διαρκούς ενημέρωσης των όσων εργάζονται σε αυτό το τομέα και εσείς Πρόεδρε θυμήσατε τη δραστηριότητα της Ευρωπόλ. Η Europol προσφατά έχει ασχοληθεί μέσω των αστυνομικών της ερευνών με το θέμα της παραχάραξης στο Darknet. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να αποτελέσει τμήμα αυτής της μόνιμης ενημέρωσης που καταφέρνει να έχει ε, ε, το οργανωμένο έγκλημα ε, και πώς θα βρούμε μέτρα τα οποία όλο ένα και περισσότερο θα αυξάνουν την αντίσταση στην εγκληματικότητα αλλά και το επίπεδο προστασίας. Γι' αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος Περικλής θα πρέπει να τονίσουμε την ανάπτυξη νέων ε, ε, πλατφορμών ανταλλαγής στο ε, Darknet. Εδώ ο εισηγητής σωστά υπογράμμισε ότι και για το θέμα του ελέγχου των χρηματοδοτήσεων. Μια άλλη πτυχή είναι ακριβώς η ευθυγράμμιση των διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης εντός του πολύετούς ε, δημοσιονομικού προγράμματος υπό τη μορφή ε, εξουσιών και ε, κατεξουδότηση πράξεων. Το πρόγραμμα που τώρα παρουσιάζει ο συνάδελφος Βιώτη δεν είναι πολύ καλά ξεκαθαρισμένο σύμφωνα με ποια βάση δηλαδή θα οριστούν οι, τα ετήσια προγράμματα. Το άρθρο 10 που αναφέρεται σε αυτά δεν ορίζεται αν θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να οριστούν με, με κατεξοδότηση πράξης ή όχι ή με εφαρμοστικές πράξεις. Τα κριτήρια λοιπόν δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα και θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο αυτά θα αριθμιστούν με κατεξοδότηση πράξη ή όχι. Επαναλαμβάνω λοιπόν την μεγάλη σημασία και το θετικό χαρακτήρα του προγράμματος και εγώ με τις τροπολογίες μου θα προσπαθήσω να συμβάλλω το έργο του συναδέλφου Dennis De Jong, τον οποίο ευχαριστώ και πάλι, όπως ευχαριστώ και την Κομισιόν για την εισήγησή της. Ευχαριστώ Κατερίνα. Αυτό ήταν το τελευταίο μας σημείο για σήμερα, οπότε κλείνουμε τώρα τη συναντρίασή μας ε, λίγο νωρίτερα. Θέλετε να ζητήσω την Κομισιόν να απαντήσει, κύριε De Γιόγκ. Σύντομα, παρακαλώ. Κύριε Κάουφ, παρακαλώ δώστε μας μια απάντηση. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή αλλά και την κυρία Κινίτσι για τις παρατηρήσεις τους, τις Το, το μικρόφωνο σας παρακαλώ, αν θέλετε να ανάψετε. Κοιτάξτε, το έγγραφο εργασία αυτό αντικαθιστά την αξιολόγηση αντικτύπου. Πρόκειται για ένα οριζόντιο χαρακτηριστικό για περισσότερα προγράμματα με περιορισμένο προϋπολογισμό. Και έχουμε ακριβώς ε, μία αναθεώρηση για να αξιολογούμε ακριβώς ε, το σύνολο και το αποτέλεσμα του προγράμματος. Και ε, σε σχέση με τους ε, δείκτες απόδοσης και αυτοί έχουν απλοποιηθεί για να έχουμε δείκτες απλούς, μετρήσιμους ε, και έναν δείκτη που θα έχει ποιοτική φύση. Και βεβαίως ε, η ε, θα προχωρήσει στην κατάρτιση ειδικών δικτών απόδοσης εάν αποδεικτεί ότι δεν μετρούν επαρκώς ε, την απόδοση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και βεβαίως ε, και στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, είναι στο πρόγραμμα εργασία. Επίσης είμαστε σε επαφή με την Κίνα για την ε, πλαστογράφηση των ολογραμμάτων ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και να υπάρχει μια σοβαρότερη επιβολή από το Κινέζικο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και από την ε, Λαϊκή Τράπεζα της ε, Κίνας. Όσον αφορά την Europol, η Europol συμμετέχει πλήρω στο πρόγραμμα. Έχουμε την στρατηγική του Περικλέους ε, που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ΕΚΤ, Europol και Κομισιόν και η στρατηγική αυτή με βάση τις πληροφορίες, τις εμπιστευτικές της Europol μας λέει που πρέπει να δραστηριοποιηθεί το πρόγραμμα. Οπότε υπάρχει η συνεισφορά της Europol και δεύτερον η πείρα της ε, Europol ε, ακριβώ ε, κινητοποιείται και χρησιμοποιείται, υπάρχει και εκπαίδευση την οποία παρέχει σε διάφορες χώρες για να τις βοηθήσει στις έρευνές τους. Και αυτή είναι μετά η λεγόμενη τεχνική αρρωγή. Όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μας, ε, αυτό το εγκρίνει η Κοπισιόν μετά από την ενημέρωση αυτής της ε, στρατηγικής και συζητήσαμε επίσης ε, το πρόγραμμα εργασίας και την έγκρισή του με τα κράτη-μέλη. Έτσι ακριβώς ε, καταρτίζεται το πρόγραμμα εργασίας και η Κομισιόν στο παρελθόν δεν ήταν υπέρ των πράξεων ε, κατά εξουσιοδότηση. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την ΕΚΦΙΝΕ. Δεν έρχεστε τακτικά εδώ. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Τσινίτσι. Λοιπόν, πριν σηκωθείτε να φύγετε, έχει ακυρωθεί το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, η επόμενη συνεδρίαση είναι 15 Οκτωβρίου. Γεια σας.